Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να αρχίσουμε. Να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη πρώτα με την εξή αλλαγή. Στο σημείο 4 είναι ανταλλαγή απόψεων την έκθεση του κ. Μπόνη αφορά το μέσο ευρωπαϊκών αξιών για να στηρίξουμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που αγωνίζονται για τις ευρωπαϊκές αξίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στις 9 ή τέλο πάντων μόλις ολοκληρώσουμε με τον κύριο Τίμερμαντς. Εντάξει, δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Ωραία, εγκρίνεται. Κροατικά, δανέζικα, λετονικά, εγγέλικ δεν θα τα έχουμε σήμερα δυστυχώ. Μα ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Έχουμε αυτά τα δύο σημαντικά λοιπόν ζητήματα και το πρώτο είναι ο διαρθρωμένος διάλογος με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Τίμερμαντς. Ο Φρανς Τίμερμαντς είναι εδώ για να συζητήσουμε το πρόγραμμα εργασιών του 2018. Αλλά βέβαια έχουμε και ευαίσθητα ζητήματα που έχουν προκύψει. Όπως γνωρίζετε, σε σχέση με την Πολωνία, την Μάλτα και πιο πρόσφατα την Σλοβακία. Οπότε θα ακούσουμε τον Επίτροπο να μας αναλύσει κάπως τις τελευταίες εξελίξεις σε αυτά τα τρία μέτωπα. Και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους συναδέρφους για να συζητήσουμε. Έχουμε χρόνο για τη συζήτηση μέχρι τις 9 με τον κύριο Τίμερμανς. Λοιπόν, ας ακούσουμε τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φρανς, καλώς ήρθατε. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Κλοντ. Και επιτρέψτε μου, παρακαλώ, πριν μπω στην ε, ουσία των θεμάτων που θα αναπτύξω, επιτρέψτε μου να σας πω ότι παρακολουθώ από κοντά την δήλωση της ε, Πρωθυπουργού Τερέσα Μέη σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων σχετικά με την ε, επίθεση ε, που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από ό,τι άκουσα από την Πρωθυπουργό Μέη, χρησιμοποιήθηκε το αέριο αυτό κατά δύο πολιτών που ζουνε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ένα αέριο ε, νευρών το οποίο απαγορεύεται Ζήτησε διευκρινήσεις η Τερέσα Μέη. Ζήτησε διευκρινήσεις από τις ρωσικές αρχές για το κατά πόσο επίτηδες χρησιμοποιήθηκε έτσι το αέριο αυτό νεύρων ή διέφυγε με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, ε, νιώθω μεγάλη αλληλεγγύη με το Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτό και με όλους μας για να υποστηρίξουμε τις βασικές μας αξίες, ε, τους ανθρώπους που ζουν στην επικράτειά μας, πρέπει να είμαστε ενωμένοι απέναντι σε μια ιδιαίτερα περίπλοκη κατάσταση με μια χώρα που βρίσκεται κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά που δημιουργεί τόσα προβλήματα με τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι βασικό για τη δικιά σας Επιτροπή. Το 2006 το Ρωσικό Κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο που επιτρέπει, είναι νόμιμο λέει, να ε, δολοφονούνται προδότες στο εξωτερικό. Αν μιλάμε λοιπόν για κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πολλά να συζητήσουμε, αλλά ας είμαστε ενωμένοι και ας εκφράσουμε όλοι μαζί την αλληλεγγύη μας απέναντι στο Βρετανικό λαό και τη Βρετανική κυβέρνηση αυτές τις δύσκολες στιγμές. Επίσης θέλω να πω ξεκάθαρα ότι εκφράζω και την ευγνωμοσύνη μου στην Επιτροπή σας και για το σκληρό έργο που έχετε κάνει, για πολλά λεπτά ζητήματα και δύσκολα, αλλά και γιατί εμένετε στο κράτος δικαίου που καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που είναι και μας αυτό που είμαστε. Πιστεύω ειλικρινά ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να εξυπηρετήσει κανείς. Ζούμε σε καιρούς που δυστυχώς πρέπει κανείς να υψώνει τη φωνή του, να επιλέγει η πλευρά. Θα σας μιλήσω λοιπόν για το κράτος δικαίου, για την Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Πολωνία, τη Μάλτα και μετά βέβαια θα είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ σε ερωτήσεις σας. Πρώτα απ' όλα για το κράτος δικαίου γενικά. Όπως ε, ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα εργασιών του 2018 θα παρουσιάσουμε πρωτοβουλία για να ενισχύσουμε το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αργότερα μέσα σε αυτή τη χρονιά με το ψήφισμα του Οκτωβρίου Ακριβώ αυτό είστε και εσεί. Σε αυτήν τη συζήτηση λοιπόν, πριν από 4-5 χρόνια ε, φαινόταν ότι δεν συζητάγαμε για θέματα κράτους δικαίου. Τώρα συζητάμε θεμελιώδεις ελευθερίες όπως συζητούσαμε για τα ψάρια ή για τα οικονομικά. Θα πείτε δυστυχώ. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει κάτι θετικό γιατί αυτό δείχνει τη δύναμή μας, ότι ακριβώ μπορούμε να συζητάμε τέτοια θέματα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα μάλιστα ακόμα και στο Συμβούλιο, όπου τα κράτη-μέλη δεν κρύβονται πια από τις ε, ευθύνε τους. Οπότε το άρθρο 2 μπαίνει στο τραπέζι. Και αυτό είναι θετικό, γιατί τελικά είναι θέμα υπαρξιακό που πρέπει να θέσουμε στους αυτούς μας. Τι Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε Πιο συγκεκριμένα τώρα για την ε, Πολωνία. Ευχαριστώ την ε, Επιτροπή σας που δεσμεύτηκε υπέρ του κράτους δικαίου στην Πολωνία και που στήριξε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα. Δεν ήταν πάντα εύκολα τα πράγματα τα τελευταία δύο χρόνια, όμως είμαι περήφανος που μπορώ να πω ότι με τον πρόεδρο Γιούνκερ, τους συνεργάτες του και ολόκληρο το Σώμα των Επιτρόπων καταφέραμε να προχωρήσουμε και να ζητήσουμε από την Πολωνία να έρθει στο τραπέζι για διάλογο. Και αυτό θέλω να το τονίσω. Υπάρχουν ε, μερικοί που θέλουν να παρουσιάσουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διχασμένη. Ότι δεν συμφωνώ με τον πρόεδρο Γιούγκερ. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μην έχετε ψευδεστήσει. θα σας απογοτεύσουμε. Ο πρόεδρος Γιούγκερ και εγώ είμαστε ακριβώ στην ίδια γραμμή σκέψη. αγωνιζόμαστε για τι ίδιε αξίε και τι ίδιε αρχέ. Και το έχουμε κάνει αυτό τα δύο τελευταία χρόνια. Εμείς ε, ε, τίνουμε χείρα προς την Πολωνία. Το κάναμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και το κάναμε να ενεργοποιήσουμε το άρθρο 7. Όχι για κυρώσει, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι ως στοματοφύλακε των συνθηκών έρχεται κάποια στιγμή όπου πρέπει κανεί να βάζει τη διαχωριστική γραμμή. Και το Κοινοβούλιο μα στήριξε γιατί στηρίζει το κράτο δικαίου. Το ψήφισμα τη 1 η Μαρτίου, το δικό σα, με ευρία στήριξη από τι πολιτικέ ομάδε, στέλνει ένα σαφέ μήνυμα ότι υπάρχει κίνδυνος ε, παραβίαση του κράτου δικαίου στην Πολωνία και γι' αυτό επήγε να δραστηριοποιηθούμε. Οπότε αποφασίσαμε να ενεργοποιήσουμε τα άρθρα 7 και συγχρόνως μπήκαμε και στην τέταρτη σύσταση για να βοηθήσουμε την Πολωνία να λύσει τα προβλήματα τα οποία εντοπίστηκαν. Έτσι λοιπόν αναφέρονται σύσταση, σε αυτή τη βήματα μπορεί να πάρει η πολωνική κυβέρνηση για να λύσει το ζήτημα. Η Κομισιόν πιστεύει ότι η πολωνική κυβέρνηση πρέπει να ανταποκριθεί σε πέντε ανησυχίες. Και θα σας τις αναφέρω όλες, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια το έκανε. σω να μην ήσασταν όλοι παρόντες, οπότε θα σας τα ξαναπώ. Πρώτον, δημοσίευση της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου της 26ης. Υπό το κράτος δικαίου καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να αποφασίζει ποιες αποφάσεις δημοσιεύονται και ποιες όχι. Εφόσον μάλιστα η δημοσίευση σημαίνει ότι μόνο τότε είναι έγκυρη μία απόφαση. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αποφασίζει τι θα δημοσιευτεί, άρα θα ισχύσει και τι όχι. Αν ασφάλει το δικαστήριο, κάποιο άλλο δικαστήριο μπορεί να το διορθώσει. Δεν είναι η κυβέρνηση όμως που θα το κάνει αυτό. Δεύτερον, ε, επαναφέροντας την ανεξαρτησία του Συνταγματικού Δικαστηρίου, φροντίζοντας να οριστούν εκείνοι οι οποίοι εγκρίθηκαν από την προηγούμενη βολή. Έπειτα, δεν πρέπει να υπάρξει μείωση της ηλικία ε, και άρα πάυση το καθηκό των διαφόρων τακτικών δικαστών. Από ό,τι φαίνεται, πολλοί θα χρειαστεί να σταξιδοτηθούν με τη ρύθμιση αυτή. Επίσης, οι δικαστές οι οποίοι ε, θέλουν να μείνουν, η κυβέρνηση αποφασίζει ότι πρέπει να απομακρυνθούν. Γιατί υπάρχει μια έκτακτη διαδικασία ε, έθεσης και πρέπει να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι μόνο γιατί υπάρχουν νέα ζητήματα, αλλά υπάρχουν ε, και διαφορετικές νομικές ρυθμίσεις. Εδώ σας παραπέμπω στην έκθεσή της Επιτροπής της Βενετίας που εξηγεί γιατί όλα αυτά είναι σε βάρος του κράτους δικαίου. Τέταρτο, τροποποιώντα ε, την νομοθεσία για τα τακτικά δικαστήρια για να αλλάξει ακριβώ ε, και η νομοθεσία ε, όσον αφορά τη συνταξιδότηση των ε, τακτικών δικαστών και την δυνατότητα της κυβέρνησης να αποφασίζει ή όχι την παράταση ε, των δραστηριοτήτων τους. Επίσης, για την ε, πάυση ακριβώ των τακτικών δικαστηρίων του, δικαστικού, του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου, που κανονικά εκλέγονται από άλλους δικαστές και όχι από πολιτικούς. Επίσης, η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε βάρος της Πολωνίας για παραβίαση ε, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα τακτικά δικαστήρια. Υπάρχει απόφαση της 27ης Φεβρουαρίου C6416 όπου αναφέρει το άρθρο 2 και 19 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέγοντας ότι σε εθνικό επίπεδο πρέπει να διασφαλίζεται η, ως ανεξάρτητη αρχή το δικαστικό σώμα, η δικαιοσύνη. Και άρα υπάρχει βάση για διάλογο με την πολιτική κυβέρνηση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Κοιτάξτε τι. Τώρα τον Ιανουάριο που μας πέρασε υπήρξαν ανταλλαγέ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Πολωνικής Κυβέρνησης ευτυχώς και συνεχίζονται σε διάφορα επίπεδα τον μήνα που μας πέρασε, την πέμπτη που μας πέρασε, ο πρόεδρος Γιούνκερ και εγώ συναντηθήκαμε με τον κύριο Μοσχαβιέτσι, τον πρωθυπουργό της Πολωνίας και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο συναντηθήκαμε και με τον Υπουργό Εξωτερικών και συμφωνήσαμε να συνεχιστεί και στη Βασοβία και στις Βρυξέλλες αυτός ο διάλογος. Επιπλέον, η Επίτροπος Γιούροβα συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών έγιναν αλλαγέ σε τεχνικό επίπεδο επίση. Οι συναντήσει αυτές έγιναν σε ένα καλό κλίμα. Ο διάλογος λοιπόν υπάρχει, αλλά ο διάλογος πρέπει να οδηγήσει και σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό προσπαθούμε τώρα. Να είσαστε σίγουροι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώνει τακτικά και πλήρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για οτιδήποτε συμβαίνει. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω ότι θα μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα αυτά ζητήματα, όπω έχει κάνει και κατά το παρελθόν. Η συνεργασία μεταξύ μα ενισχύει τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οδηγεί και το Συμβούλιο να αναλάβει πρωτοβουλίε για να λύσει αυτά τα ζητήματα. Οπότε σα είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων. Πριν να περάσω στη Μάλτα, επιτρέψετε μου να αναφερθώ στις δολοφονίες δημοσιογράφων στη Μάλτα και στην Σλοβακία. Η Επιτροπή δίνει τεράστια σημασία στον πλουραλισμό και την ελευθερία του λόγου. Η δολοφονία, ο εκφοβισμό δημοσιογράφων είναι κάτι που δεν έχει θέση ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε σε οποιαδήποτε δημοκρατία. Οπότε καταδικάζουμε τη δολοφονία του Γιάννη Κουτσιακ και τη συντρόφου του τον προηγούμενο μήνα, όπω επίση και τη δολοφονία τη Μαλτέζα δημοσιογράφου στη Μάλτα είναι κάτι το οποίο έχει σοκάρει ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινότητα. Και όταν μιλάω για ευρωπαϊκή κοινότητα εννοώ τις ευρωπαϊκές κοινωνίε. Είναι κάτι που δεν περιμέναμε ποτέ να συμβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι όμως που συμβαίνει ότι υπάρχει τρόπος να εκφοβιστούν οι δημοσιογράφοι και να κάνει κανείς τη ζωή τους πιο δύσκολη και τη δουλειά του πιο δύσκολη. Και αυτό αντιβαίνει στο κράτο δικαίου. Όπω έχουμε πει ξανά και ξανά στην περίπτωση τη Πολωνία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένει σε βάθο έρευνα από τι αρχέ για τον θάνατο τη δάφνη Γαλλίσια και χαιρόμαστε για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, Όμω θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τι αρμόδιε αρχέ να πιέσουν να ολοκληρωθεί η έρευνα με ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για την περίπτωση της ε, Σλοβακίας. Δεν πρέπει να μείνει ε, καμιά πέτρα χωρίς να την ε, σηκώσουμε για να ψάξουμε και να αποδοθεί έτσι δικαιοσύνη. Εδώ βλέπετε στην περίπτωση της Σλοβακίας, δεν πρόκειται μόνο για το ποιος ε, πυροβόλησε, ε, πρόκειται και για το ποιος έβαλε κάποιον να πυροβολήσει. Το ίδιο ισχύει και για τη Σλοβακία και για την Μάλτα, δηλαδή θέλουμε να βρούμε από πού ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Και ό,τι επεκτάσεις και αν έχει αυτό το ζήτημα πρέπει να πάμε προς κάθε κατεύθυνση χωρίς καμία επιφύλαξη. Για τη Μάλτα τώρα πιο συγκεκριμένα. Σημείωσα ότι συζητήσατε με την συνάδελφό μου Γιούροβα που είναι αρμόδια για πολλά από αυτά τα ζητήματα. Εμείς χαιρόμαστε πάντως για την έκθεση της Αντόκ ε, Αποστολής που πήγε υπό την κυρία Γκόμες στη Μάλτα. Και σημειώσαμε όλα όσα αναφέρετε στην έκθεσή σας. Παρακολουθούμε και εμείς όλες τις πτυχές που είναι της αρμοδιότητάς μας και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να τηρείται πλήρως. Επιμείναμε και επιμένουμε στι Μαλτέζικες αρχές να πιέσουν με τη σειρά τους ώστε να αντιμετωπιστούν όλες οι ανησυχίες. Σε αυτά τα πλαίσια χαίρομαι για την ανακοίνωση του Υπουργού Δικαιοσύνη της Μάλτας που λέει ότι θα κοινοποιήσει η Μάλτα πολύ σύντομα την πρόθεσή της να συμμετάσχει και αυτή στην υπηρεσία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Είναι κάτι πολύ θετικό αυτό. Αλλά δεν θα σταματήσουμε εκεί. Επιμένουμε. Οι Μαλτέζικε Αρχέ πρέπει να συνεχίσουν να πιέζουν προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλε οι ανησυχίε που υπάρχουν. Και αυτό πρέπει να γίνει με επιτυχία, με διαφάνεια, έτσι ώστε να πάψουμε να έχουμε ανησυχίες εμείς, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και η κοινωνία στο σύνολό της. Όσον αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την νομοποίηση παρανομού χρήματος. Το ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα ακριβώς προσπαθεί αυτό να αποφύγει και είναι ζωτική σημασία να το πετύχουμε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει οδηγία πλαίσιο που αλλάζει. Η Επιτροπή παρακολουθεί πώς ενσωματώνονται οι νέοι κανόνες Στι 3 Ιανουαρίου που μας πέρασε κοινοποίησε η Μάλτα ότι ενσωμάτωση νομοθεσία της στην ε, τρίτη οδηγία για την ε, ε, καταπολέμηση της νομιμοποίηση παράνομου χρήματο. Αξιολογούμε τώρα τις διατάξεις. Τις εκτιμούμε. Αλλά μας ενδιαφέρει βέβαια και εφαρμογή. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σε ανάλυση για τις νομικές πτυχές και τις τεχνικές πτυχές βλέπουμε προς το παρόν ότι δεν υπάρχει, δεν έχει εντοπιστεί συστηματική παραβίαση της νομοθεσίας αυτής, όμως παραμένουν σοβαρά ερωτήματα για το πώς εφαρμόζονται από τις αρμόδιες αρχές αυτές οι διατάξεις και πώς ενημερώνεται το κοινό, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται για να έχει εμπιστοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν συνεχίζει να ζητάει πληροφορίες απευθείας από τις αρχές και ζητά επίσης από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή να εκτιμήσει κατά πόσο οι τραπεζικοί επόπτες είναι εξοπλισμένοι με ό,τι χρειάζεται για να φέρουν σε πέρα στα καθήκοντά τους και κατά πόσο οι οικονομικές αρχές της Μάλτας φέρουν σε πέρα στις δικές τους αρμοδιότητες, εποπτείες κτλ. Ε, παρόλο που δεν έχει υπάρξει δράση κατά της τράπεζας πιλάτες και άλλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης παρακολουθεί από κοντά την ε, αξιολόγηση της ε, νομοθεσίας της Μάλτας και να ξέρετε ότι και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει βοηθήσει πολύ, γιατί και εκείνοι αναλαμβάνουν την ευθύνη, παίρνουν πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα και τους ευχαριστώ ενώπιόν σας. Όσον αφορά τώρα την ε, ανταλλαγή, δηλαδή την απόδοση της ηθαγένειας της Μάλτας έναντι επενδύσεων. Και εδώ παρακολουθούμε την νομοθεσία και την πρακτική και δίνουμε κατευθυντήριες γραμμέ στις χώρε μέλη. Υπάρχει έρευνα για να προετοιμάσουμε τη σχετική μας έκθεση για το 2018, οπότε βλέπουμε στην πράξη πώς εφαρμόζεται το πρόγραμμα αυτό στις διάφορες χώρες. Και θέλω εδώ να τονίσω το ψήφισμα της 14 ης Νοεμβρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το κράτο δικαίου στη Μάλτα και τις συστάσεις που συμπεριλαμβάνει η κοινή ε, αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της δικιάς σας Επιτροπής και της Επιτροπής ΠΑΝΑ. Όλα αυτά δείχνουν τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι το οποίο μας βοηθάει εμάς όλους ιδιαίτερος, γιατί κάνει το έργο μας πιο εύκολο και μπορούμε έτσι να δουλέψουμε περισσότερο σε βάθος. Σας ευχαριστώ. Τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν βέβαια τα δικά τους προνόμια, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, συνεργάζονται και μεταξύ τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το απαιτεί αυτό. Στα πλαίσια ερευνών μπορεί να αποδοθεί η ηθαγένεια βάσει μιας αυθεντικής σχέσης του ετούντος με τη χώρα. Και αυτό μετά από ένα εύλογο διάστημα όπου κατοικεί στη χώρα ο ενδιαφερόμενος. Η Μάλτα λοιπόν συζήτησε ήδη από τον Ιανουάριο του 2014 το πρόγραμμα αυτό και εμείς επιμείναμε ότι πρέπει να μπορεί να αποδείξει ο ετόνο την στενή σχέση που έχει με τη χώρα και ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατοικίας του στη χώρα. Επιμένω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη την διαφθορά και πρέπει να προλάβουμε τη διαφθορά, κάτι το οποίο είναι προτεραιότητα και περιλαμβάνεται και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η έκθεση βάσει του εξαμήνου για τη Μάλτα αναφέρει την καταπολέμηση της διαφθοράς και λέει ότι η διαφθορά αποτελεί ένα προβληματικό παράγοντα στην Μάλτα και σημειώνει το κατακαιρματισμένο τοπίο των διαφόρων αρχών και υπηρεσιών που ασχολούνται με τη διαφθορά στην Μάλτα. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση και είναι η προτεραιότητά μας. Μας ενθαρρύνουν και οι Μαλτέζικε αρχέ με την απόφασή του να ενταχθεί η χώρα στην υπηρεσία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Ρουμανία τώρα. Πήγα την 1η Μαρτίου στο Βουκουρέστι για να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα για συνεργασία και παρήθευση και το σύστημα του σχετικό του CVM. Πώ να ξεπεράσουμε τα επίμαχα ζητήματα όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα και τη φορολόγηση του δικαστικού τομέα. Στόχο μου Θέλω η μεταρρύθμιση να επανέλθει στην κανονική πορεία. Μετά την επίσκεψή μου, παρέμεινε επιφυλακτικά αισιόδοξο η δυνατότητα να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Όμω, πρέπει να δεχτούμε ότι απομένουν δυσκολίες, κυρίω δοθήσει της πολλώσεως των θέσεων των πολιτικών και του δικαστικού κλάδου. Σε σχέση με το CVM, λοιπόν, το συνέκρινα με ένα μαραθώνιο. Η Ρουμανία είναι στην τελική ευθεία του μαραθωνίου είναι σημαντικό να συνεχίσει κανείς να τα έχει σωστή κατεύθυνση και όχι από την άλλη μεριά. Έδωσε σαφές μήνυμα. Πριν φτάσεις στον τερματισμό δεν αλλάζεις πορεία. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε. Όμως η Ρουμανία έχει τελική ευθύνη και οι αρχές της. Ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ είπε σαφώς ότι επιθυμεί να λήξει το CVM κατά τη διάρκεια αυτής της ζητίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή είναι η φιλοδοξία μου. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Αυτό δεν αποτελεί προθεσμία. Μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν οι συστάσεις ακολουθηθούν. Είναι εφικτό, είναι εφικτό. Αλλά πρέπει να συνεχίσει η προσπάθεια με αποφασιστικότητα, όπως και πριν. Και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από αυτή που είδαμε τον τελευταίο χρόνο. Χρειαζόμαστε στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμών της Ρουμανίας. Η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να τερματιστεί η τεχνογνωσία τη Επιτροπή Βενετία και τη Επιτροπή Γκρέκο πρέπει να γίνει σεβαστή. Είναι εμπειρογνώμονε αυτοί με μεγάλο. την χάνουν μεγάλου σεβασμού. Λοιπόν, να κλείσω λέγοντα ότι το κράτο δικαίου και το σεβασμό ε, των θεσμών δεν μπορεί να τον βάλει σε κανόνες και μόνο. Είναι θέμα πολιτική νοοτροπία. και αλληλεπιθέσει μεταξύ θεσμών δημιουργεί πολιτική νοοτροπία κακή για το κράτος δικαίου. Οπότε η παραπληροφόρηση κατά των δικαστών είναι κάτι κακό για το κράτος δικαίου. χρηματοδότηση επιγραφών που κατηγορεί τους δικαστές που λέει ότι είναι κομμουνιστές διαφθαρμένοι είναι κακό για το κράτος δικαίου. Και είναι και κακό για την πραγματικότητα, διότι αυτά δεν είναι αληθή. Δεν μπορεί ο ένας θεσμός να κυνηγάει τον άλλον. Παρομοίως, οι δικαστικοί θεσμοί δεν θα πρέπει να διώκουν το κοινοβούλιο την κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός των θεσμών και την διάκριση των εξουσιών. Έτσι λειτουργεί η κατάσταση, σωστά. Λοιπόν, χρειάζεται μια ανατροπή που πρέπει να λυγηθεί για το δικαίου μέσω παιδείας. Ξεχνάμε την παιδεία, την εκπαίδευση. Το είπα και στην αρχή. Και είναι η τελευταία μου κουβέντα αυτή, πριν να απαντήσω σε ερωτήσεις. Είμαστε πλέον ευάλωτοι από ό,τι θεωρούμε δεν είναι κάτι το οποίο είναι άθραυστο που έχουμε στα χέρια μας. Καμιά φορά εμείς χειρότεροι αυτού που θεωρούμε. Πρέπει όμως να μιλάμε, να εκφράζουμε αυτά που θέλουμε και έτσι να ενισχύσουμε το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ας ακούσουμε τα μέλη. Συνάδελφοι, Όλοι οι παρόντες θέλουν να μιλήσουν. Σας παρακαλώ, περιοριστείτε σε ένα δίλεπτο. Αν έχουμε χρόνο στο τέλος, θα κάνουμε κι άλλο γύρο. Ίσως να υπάρχουν και κάποιοι θέλουν να δευτερολογήσουν. Είναι πολύ σημαντικά θέματα αυτά. Και ασχολούμαστε με αυτές τις χώρες που αναφέρθηκαν. Ένα δίλεπτο στην αρχή και αν περισσέψει χρόνος θα ακούσουν ερωτήσει. Η κυρία Ματσόλα έχει το λόγο για το έλεγχο. Ευχαριστώ, Κλοντ. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε Τίμερμαντ. Υπήρξατε σαφέστατος. Ό,τι και να σκέφτονται οι πρωθυπουργοί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν είναι η τυραννία της πλειοψηφίας η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι η κυβέρνηση κυβέρνηση μας ψηφία με τα δικαιώματα της απόλυτης πλειοψηφίας. Αυτά είναι άρρηκτα συνδεμένα. Και η διαφθορά με ατιμορρησία σκοτώνει τα δικαιώματα. Άρα είναι ασύμβατη με τη λειτουργία του κράτου δικαίου γι' αυτό. Χρειαζόμαστε ανεξάρτητο δικαστικό κλάδο. Δεν θα επηρεάζεται από πολιτική επιρροή και επί χάρτου και στην πράξη. Χρειαζόμαστε ελεύθερα και προστατευμένα ΜΜΕ και ελευθερία του λόγου. Γι' αυτό θέλουμε να διαφυλαχθεί το κατοσδικαίο δημοκρατία και τα δικαιώματα των ε, πολιτών στη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και παντού στην Ένωση. Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι που δολοφονήθηκαν, δολοφονήθηκαν πριν ε, σε μια απόσταση πέντε μέρες. Η Δάφνη στη Μάλτα και οι άλλοι στην ε, ε, Σλοβακία προσπαθούσαν να διαρευνήσουν ε, το ξέπλυμα χρήματο, τη μαφία κλπ. Δεν είναι απλώ δύο δολοφονίες, αλλά είναι τα διάφορα θέματα που κρύβουν. Η εκτέλεση αυτών των δημοσιογράφων εξέθεσε τα προβλήματα. Όπου και να ρίξουμε τη ματιά μα, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κενό μεταξύ των προσδοκομένων δικαιωμάτων των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και των μηχανισμών που είναι διαθέσιμοι για να εξασφαλίζουν την προστασία. Γι' αυτό αυτό το κοινοβούλιο και ένα μηχανισμό ευρωπαϊκό που προστατεύει τη δημοκρατία και το κάτω δικαίου και τα μελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών σε όλα τα κράτη-μέλη είναι πολύ σημαντικά. Αυτό θα συμπεριλάμβανε συγκεκριμένα μέτρα που θα προστατεύουν διώξει και μηνύσει που ασκούν πιέσει στου δημοσιογράφου και στι ΜΚΟ. Υπό πολλέ μορφέ μπορεί να υπάρχει ο μηχανισμό. Ετήσια αξιολόγηση, είπαμε το χάρη, με συστάσει για κάθε κράτο μέλο. Να συνδυάζει σειρά εκθέσεων κατά χώρα. Δεν είναι κάτι καινόφανε. Κάθε κράτο μέλο θα υπόκειται στον ίδιο έλεγχο. Μέσω ανεξάρτητου φορέα ελέγχου που θα εξετάζει λεπτομερώς ποια είναι η κατάσταση σε κάθε χώρα. Δεν μας ενδιαφέρει να κυνηγήσουμε μια χώρα, Θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα. Λοιπόν, βάσει των όσων είπατε στην αρχή, και σε ευχαριστούμε γι' αυτό, ρωτώ λοιπόν, υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του μηχανισμού. Βέβαια, στον παρόδοτε, έχετε πλήρη υποστήριξη κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Κύριε Τσίπελ, S&D. Σα ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι δεν δείχνει θέμα. Η ανεξαρτησία η ανεξάρτητα, τα ανεξάρτητα λοιπόν μέσα ενημέρωση και τα επιδευτικά κράτη-μέλη μέσα ενημέρωση αποτελούν προδιαγραφή για το κράτο δικαίου. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε και οι δύο οι δημοσιογράφοι ερευνούσαν περιπτώσει διαφθορά, ερευνούσαν διαπλοκέ μεταξύ εγκλήματο και πολιτική. Αυτό ανησυχεί λοιπόν όλου μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι καλό που όλοι μαζί αναζητούμε και στις χώρες αυτές, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσπαθούμε λοιπόν να αντιπιστώσουμε ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά. Γιατί μόνο έτσι θα βρούμε και το τι μπορεί να γίνει για να επιληθεί η κατάσταση. Και χαίρομαι ιδιαίτερω που ο Υπουργό Ιστορικών στη Σλοβακία αποσύρθηκε από τα καθήκοντά του για να δώσει μία κάποια πολιτική και ηθική, αν θέλετε, ε, συνέχεια και να αναλάβει τέτοιε ευθύνε. Ε, δεν αρκεί βέβαια αυτό ένας από τους λόγους ε, των όσων ε, είδαμε τον τελευταίο μήνα είναι η διαφθορά. Αν ισχύει αυτό, θα πρέπει η διαφθορά λοιπόν να δραματιστεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Πέρα λοιπόν από το τι μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε τις έρευνες στην ε, Μαλτά, στην Σλοβακία, θα ήθελα να θίξω και το θέμα των διαφόρων ερευνών σε ό,τι αφορά και διαφορών αναφορών σε ό,τι αφορά την ε, διαφθορά στην ε, Ουγγαρία. Τι μπορούμε να κάνουμε εκεί για να σταματήσουμε τα περιστατικά διαφθοράς και να επηρεάσουμε την κυβέρνηση. Θα ήθελα να επίση να ξέρω στο πλαίσιο αυτό κατά πόσο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να υποστηρίξει αιτήματα για να αλλάξουν οι κανόνε για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό να μπει μια αλφαρεσιμότητα για τη χορήγηση ευρωπαϊκών πόρων σε άλλες χώρες σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Πέραν τούτου, να θέσω και το θέμα της Πολωνίας. Χαίρομαι ιδιαίτερω και υποστηρίζουμε το γεγονός ότι επικαλείται το άρθρο 7, 7.1 συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να περάσει στο 7.2. Δεν ξέρουμε όμως ποια θα είναι οι αντιδράσεις της Πολωνίας στους κόλπους του Συμβουλίου. Πείτε μας δύο λόγια. Θα μας βοηθούσε. Κατά πόσον ε, αναμένεται κάποια υποστήριξη μέχρι το Μάρτιο. Και πέραν τούτου, πέρα από τα όσα ισχύουν στα πλαίσια του Α7, να θέσω και πάλι το θέμα μιας νομικής πράξης η οποία έχει αποφασιστεί τον Δεκέμβρη του 2016, όπου Ω τελευταίο σημείο αναφέρεται ότι υπό τον όρο αυτό τα δικαιώματα συνταξιοδότησης αφαιρούνται από όλους τους αξιωματούχους και τις οικογένειές τους, ακόμα και αν πρόκειται για μία ημέρα. Πώς ε, λοιπόν θέλετε την κατάσταση αυτή, σας παρακαλώ να δείτε το χρονικό όριο, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Γιούρεκ από πλευρά των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, την ευγνωμοσύνη μου προς τον κύριο Τίμερμανς που είναι μαζί μας σήμερα. Είπατε ότι θα έχουμε ευκαιρία να κάνουμε και μια πιο γενική συζήτηση, όχι μόνο να επικεντρωθούμε σε μεμονωμένες χώρες. Χαίρομαι λοιπόν που γίνεται αυτή η γενική συζήτηση σήμερα θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια θέματα τα οποία αναφέρατε και τα οποία θίξατε. Κάποιοι ζήτησαν ε, την εκτίμησή σας ό,τι αφορά το νόμο για την ευθανασία στις κάτω χώρες. Βάσει και της παρουσίασης ε, των θεμάτων αυτών από την εφημερίδα του ε, Μιλάμε για την περίπτωση μιας γυναίκας η οποία ήταν ε, στο νοσοκομείο και τελικά την άφησαν να πεθάνει παρά τη θέλησή της. Ε, ε, σας έστειλα το αίτημα αυτό και έλαβα μία απάντηση η οποία έλεγε δεν αντιμετωπίζουν, δεν ε, πραγματευόμαστε θέματα ευθανασίας. Δεν ρώτησα για την ευθανασία, μίλησα για τα δικαιώματα ενός ανθρώπου. Ένα ανθρώπου ο οποίος θανατώθηκε χωρίς να το επιθυμεί και ήθελα να ξέρω κατά πόσον υπάρχει ανοιχτό πνεύμα για τα θέματα αυτά. Πριν από κάποιο καιρό είπατε ότι αυτά είναι fake news, είναι ψεύτικες ειδήσει. Δεν είναι ψεύτικες ειδήσει. Να μην μιλάμε όμως για ψεύτικη, ψεύτικο κράτο δικαίου. Ε, και επίση να δούμε πώ εκτιμάται και το γαλλικό δίκαιο που επιτρέπει δύο έτη φυλάκισης αν υπάρχει τέτοιο θέμα ηθικής πίεσης όπως αποκαλείται κατά ενός ατόμου. Δεν έχουμε πολλά χρόνια να τα συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα, αλλά πείτε μου κάπως σύντομα ποια είναι η απάντησή σας, γιατί η απάντησή σας ε, στις αξιώσεις, στις ε, αντίθετες ε, έχουν σημασία. Και μην θεωρήσετε ότι είμαστε κατά της Ευρώπης. Απλά θέλουμε να αναφέρουμε θα ήθελα να ακούσω λοιπόν την δική σας δήλωση. Δεν είμαστε κατά της Ευρώπης, είμαστε κατά κάποιων πολιτικών και τις αμφισβητούμε. Δεν αμφισβητούμε την καλή σας θέληση. Η κυρία Βίξτρεμ για την άλλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ευχαριστήσω και σας κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμαν, που είστε μαζί μα σήμερα και πάλι. Παρά το γεγονό ότι είναι και προχωρημένη η ώρα, είναι πραγματικά κρίσιμο το ζήτημα το οποίο καλούμαστε να συζητήσουμε σήμερα και εκτιμώ όλου ιδιαίτερω το γεγονό ότι μιλάμε για κράτο δικαίου και σε ό,τι αφορά την πρόθεση μια νοοτροπία, μια κουλτούρα. Και αυτό ενδεχομένω το έχουμε παραβλέψει τελευταία. Γιατί προσπαθούμε να προστατεύσουμε, προσπαθούμε να διδάξουμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια νοοτροπία σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου και αυτό θα έπρεπε ενδεχομένω να το έχουμε προωθήσει. Ιδάλω δεν θα βλέπαμε να δολοφονούνται δημοσιογράφοι στη Μάλτα, στη Σλοβακία και όπου αλλού. Είναι πολύ ανησυχητική η κατάσταση. Σήμερα εστιζόμαστε πολύ στην Πολωνία για προφανείς ε, λόγους μετά την ε, το άρθρο 7 το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή για την Πολωνία και ξέρω ότι θα ακολουθήσει μια επίσημη απάντηση της πολωνικής κυβέρνησης στις 20 Μαρτίου προβλέπετε. Θα ήθελα να ξέρω τι θα κάνουμε στο ενδιάμεσο. Θέλετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μας για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά πιστεύω και το πιστεύω πραγματικά βαθιά ότι αν είχαμε πριν από κάποια χρόνια λάβει δράση κατά της Ουγγαρίας, δεν θα είχαμε τέτοιες συμπεριφορές ταυτόσιμες αντιγραφείς από πλευράς της Πολωνίας. Και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να καταλήγεται έτσι το κράτος δικαίου. Θα πρέπει να μπει ένα τέλος και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει κάτι ενδιάμεσο μεταξύ της ε, μηδενικής δράσης και της πυρηνικής βόμβας. Άρα, ο μηχανισμός της παρακολούθησης των κρατών μελών είναι κρίσιμη σημασία και υπάρχει ευρία υποστήριξη από πλευρά του Κοινοβουλίου προς αυτόν. Πείτε μας λοιπόν, τι προβλέπετε. Ξέρω ότι δεν ε, ενθουσιάζεστε, αλλά ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει έναν τρόπο να αποφύγουμε τέτοιε καταστάσει και σε άλλα κράτη-μέλη. Κάποιο άλλο, υπήρχε την νομίζω, δεν κάνω λάθο, η κυρία Σίπελ, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια αιρεσιμότητα, μια αμοιβαιότητα σε ό,τι αφορά την τήρηση του κράτους δικαίου και της, ε, των ευρωπαϊκών πόρων, κονδυλίων που λαμβάνει μια χώρα. Πείτε μας, αυτό θεωρείτε ότι αποτελεί μια ενταχόμενη λύση. Ευχαριστώ. Η κυρία Ένστα από την ΚΟΕ τώρα. Ε, σας ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, ακούγοντας αυτά που λέτε, εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι υποστηρικτριά σας. Σύμφωνο. Φαίνεται ότι μιλάμε για την, το μέλλον της Ευρώπης, για την διασφάλιση του πρώτου δικαίου, το μέλλον της Ευρώπης, αλλά μιλάτε και αναφέρετε τεράστιο γκάμα παραβιάσεων των ευρωπαϊκού δικαίου. Αναρωτιέμαι λοιπόν όταν τα ακούω όλα αυτά, πού έχουμε φτάσει. Θα μπορούσα να σας κάνω και μια προκλητική ερώτηση με ένα μικρό χαμόγελο. Τι ποσοστό της εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, έχει να κάνει με την ε, τήρηση του ευρωπαϊκού δικαίου από πλευρά των ευρωπαϊκών κρατών. Εν πάση περιπτώσει, θα ήταν ενδιαφέρον να το ακούσουμε αυτό. Έτσι όπω έχουν οι συνθήκε μα τώρα, έχουν εφαρμογή, έχουν εφαρμογή σε αυτά που ζούμε σήμερα, αρκούν, πρέπει να τι αλλάξουμε Τι συνθήκε. Τα βγάζει πέρα αυτό το άμυρο το άρθρο 7. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρέπει να τα ελέγξει όλα αυτά, να παρέμβει, να τα στείλει αυτά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι. Η Γερμανίδα καγκελάριο έκανε την πρόταση όχι να γίνει τροποποίηση των συνθήκων στην παρούσα φάση, αλλά μήπως τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα ευρωπαϊκά ταμεία θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε και αυτά, αν κανείς δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του σε ό,τι αφορά τους προσφύγει. Για παράδειγμα, πείτε μας ε, την άποψή σας. Ε, γιατί έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά στο θέμα αυτό. Κατά δεύτερον, φαίνεται ότι το επάγγελμα του δημοσιογράφου έχει γίνει ένα από τα πιο επικίνδυνα στον κόσμο. Μάλτα, Σλοβακία, τρέμει το φιλοκάρτη μας με αυτά που συμβαίνουν. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έμφαση, ασκεί πίεση προκειμένου να υπάρχει ανεξάρτητη διεκπεριέωση των περιπτώσεων αυτών και των ερευνών αυτών. Και τελευταία ερώτηση. Ουγγαρία. Δεν είπα τίποτα για την Ουγγαρία. Εντύπωση μου κάνει. Δεν το συνηθίζεται. Έχουμε, όπως ξέρετε, έχουμε εγκρίναμε και ένα ψήφισμα, αυτός ο νόμος κατά τον ΜΚΟ αποτελεί καταστροφή. Πώς θα το προωθήσετε και αυτό στις διαπραγματεύσει. Πείτε μας δύο λόγια. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σαρτζετίνη για το των Πρασίνων, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πράγματι, νομίζω ότι έχετε δίκιο, κύριε Τίμερμαντς, ότι έχετε δίκιο, ότι οι δημοκρατίες είναι πιο ευάλωτες από ό,τι νομίζουμε τελικά. Δεν μπορούμε βέβαια να διορθώσουμε τα ζητήματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου μόνο νομοθετώντας. Είναι και θέμα νοοτροπία, ναι. Αλλά δεν θα έπρεπε να κοιτάξουμε πώς προσεκίζουμε αυτό το ζήτημα. Είναι κακό όταν ακόμα και εσείς πάτε στην Πολωνία και εξηγείτε, λέτε σας παραπέμπω στην Επιτροπή της Βενετίας, διαβάστε τα εκεί και δείτε τα. Και εγώ που θέλω πρέπει να ασχοληθώ με την Επιτροπή Βενετίας, Λανθαρότε, την Αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Αρμόδιο ε, Απεσταλμένο κλπ. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς είναι να το μας λένε ότι πρέπει να αποταθούμε αλλού. Δηλαδή εμείς δεν δημοσιοποιούμε τις ε, διάφορες διαδικασίες επί παραβάση. Θα έπρεπε για να καταλάβουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία επιπαραβάση. Ή όταν ασχολούμαστε με τις διακρίσεις που γίνονται στην Ουγγαρία σε βάρος δικαστών και εκεί διακρίσεις που γίνανε βάση ηλικίας. Λοιπόν, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Και αυτό ε, θα έπρεπε να είναι να είμαστε ανοιχτοί, να είμαστε ειλικρινεί, με διαφάνεια να αντιμετωπίσουμε τα θέματα. Γιατί συμφωνώ με τη Σεσίλια Βίλστρομ. Αν πριν από μερικά χρόνια είχαμε ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα στην Ουγγαρία, ε, δεν θα είχαμε το copy-paste τώρα. Και ναι, είναι προβληματικό. Προχωράτε μεν με την Πολωνία, αλλά τελικά εξαρτώμεθα από τα δύο τρίτα πλειοψηφία σε αυτό εδώ το σώμα για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της Ουγγαρίας. Και τέλος, Πρόεδρε, αν στις 20 Μαρτίου δεν υπάρξει απάντηση από τους Πολωνούς, έχει εκπνεύσει δηλαδή η τρίμηνη προθεσμία, εσείς εντάξει, καλά κάνετε που δίνετε τέτοιες προθεσμίες, αλλά και δεν απαντήσουν και ούτε και οι Βούλγαροι νομίζω ότι είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν. Τι θα γίνει μετά τις 20 Μαρτίου λοιπόν, αν δεν έχει προκύψει τίποτα καινούριο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και για αυτή την ερώτηση που αναφέρεται στην εργαλειοθήκη που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τι γίνεται με τη διαδικασία του παραβάση, τι περιλαμβάνει. Ο κύριος Μπόνι τώρα. Θα μιλήσω πολωνικά. Ευχαριστώ πολύ. Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Πρώτον, για την Πολωνία, καμία από τις προσδοκίες που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, τηρηθεί τελικά. Ήρθε η ώρα για νέα δράση. Βλέπουμε νέες πρωτοβουλίες όμως από την άλλη πλευρά που παραβιάζουν τα δικαιώματα των πολιτών. Ε, παρουσίασε τη λεγόμενη Λευκή Βίβλο η πολωνική κυβέρνηση. Διαβάστε τη προσεκτικά παρακαλώ και δείτε τη διαφορά ανάμεσα στο τι είναι αλήθεια και τι είναι προπαγάνδα. Υπάρχει μια παράγραφος που λέει ότι οι δικαστές είναι κυρίως εκπρόσωποι του παλιού κομμουνιστικού συστήματος. Ξεκίνησε το 99 η αλλαγή και ο μέσος όρος ηλικίας των δικαστών είναι 41. Οπότε, δεύτερον, δολοφονίες δημοσιογράφων στη Μάλτα, στη Σλοβακία. Ποιο είναι το επόμενο βήμα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ελευθερίες παρά μόνο αν υπάρχει και ελεύθερη δημοσιογραφία. Θέλω λοιπόν να καλέσω τον Επίτροπο με στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρακολουθήσει το θέμα των ελευθεριών στην δημοσιογραφία και να κάνετε ό,τι μπορείτε για να διευκρινιστεί τελικά το τι έγινε. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε δημοκρατία και ελευθερία χωρίς δημοσιογράφους και δεν μπορούμε να έχουμε ελευθερίες και δημοσιογραφία παρά μόνο αν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν την ελευθερία να δρουν πλήρως σε όλες τις χώρες μέλη. Στη ΛΥΜΠΕ θα μιλήσουμε σε λίγο για τη χρηματοδότηση τέτοιων οργανώσεων σε τοπικό επίπεδο. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή για να τη στηρίξουμε. Θα ήθελα και ο Επίτροπος να τη στηρίξει. Τέλος, Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Ρουμανία, Μάλτα. Βουλγαρία εν μέρη. Τελικά φαίνεται ότι έχουμε μια κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε αντιμέτωποι με κρίση εδώ. Και θα χρειαστεί μια μεγάλη συζήτηση. Καλό είναι που συζητάμε για όλα αυτά τα θέματα τώρα. Πρόεδρος, ε, δυόμιση λεπτά είναι τα δύο. Καλά. Πρέπει να σας ε, διακόπτω. Εντάξει, εσείς έχετε και το κείμενό σας. Μαρτίνα Άντερσον. Ε, πώς να πω στη Μαρτίνα Άντερσον, να τηρήσετε οδήλεπτο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Δεν θα επαναλάβω αυτά που σας ρώτησαν οι προλαλήσαντες για το θέμα που μας απασχολεί, το Brexit. Θα μιλήσω για τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Όλοι γνωρίζουν εδώ ότι υπάρχουν ε, τα διάφορα κεφάλαια που προβλέπουν ε, θεμελιώδη δικαιώματα. Η Βρετανική κυβέρνηση τι είπε. Είπε ότι δεν έχει ενσωματώσει στην Εθνική Νομοθεσία τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, γιατί λέει δεν υπάρχει τίποτα καινούριο στη Χάρτα αυτή Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για να ενσωματώσει. Εμείς στη Βόρεια Ιρλανδία δεν έχουμε κυβέρνηση αυτή τη στιγμή για πολλούς λόγους και ένας από όλους είναι ότι δεν υπάρχει ισότητα. Στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ακριβώς αναφέρεται η ισότητα στη, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα περί τίνος πρόκειται, ενώ στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μιλάει για ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρέπει λοιπόν να δεχτεί τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η Βρετανική κυβέρνηση είπε ότι δεν θα μειωθούν τα δικαιώματά μας μετά το Brexit. Όμως πρέπει να διασφαλιστεί αυτό, γιατί μετά την εκστρατεία για τα δικαιώματά μας, 50 χρόνια μετά δεν είναι δυνατόν τώρα να διαπιστώσουμε ότι μειώνονται τα δικαιώματά μας. Θα έχουμε συζήτηση αύριο στην Ολομέλη για το Brexit. Πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μειωθούν τα δικαιώματά μας. Και αυτό είναι κάτι που δεν έχει να κάνει μόνο με την Βόρεια Ιρλανδία, γιατί εμείς στην ΚΟΕ έχουμε ετοιμάσει μία έκθεση για τις επιπτώσεις ε, που θα υπάρχουν στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, Βόρειας Ιρλανδίας όταν δεν θα παρεμβαίνει καθόλου η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Εμείς δεν θα έχουμε στη Βόρεια Ιρλανδία την προστασία της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ενώ οι Βρετανοί που θα ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν αυτή την προστασία. Συνεπώς, δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται η άρνηση της χάρτας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κυρίως για την Βόρεια Ιρλανδία, εμείς γι' αυτό ζητάμε να παραμείνουμε. Δεν είναι μόνο το θέμα των συνόρων με την Ιρλανδία, είναι ότι δεν θέλουμε να οπισθοχωρήσουμε, να πάμε πίσω να βρεθούμε σε ένα χώρο όπου αρνούνται τα θεμελιώδη μας δικαιώματα. Εφόσον η Χάρτα Θεμελιών Δικαιωμάτων δεν θα ισχύει στην Βόρεια Ιρλανδία, εμείς δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στο προηγούμενο καθεστώς. Ευχαριστώ πολύ, Άννα Γκόμες. Επίτροπε, σωστά τα είπατε, ότι οι πιέσεις επί των δημοσιογράφων, η δολοφονία των δημοσιογράφων και η ψυχολογική πίεση στους άλλους είναι κάτι βασικό για το κάτω στικαίο. Τι βλέπουμε και στη Μάλτα και στη Σλοβακία με αυτές τις αποτρόπες δολοφονίες ότι υπάρχει ένα κοινό στοιχείο. Η εμπλοκή της μαφίας, του οργανωμένου εγκλήματος και αποκάλυψη, ε, εμπλοκή ανθρώπων που είναι στην εξουσία ε, και προσπαθούν να αποκαλύψουν δημοσιογράφοι και δολοφονούνται για να εμποδιστεί η αποκάλυψη. Πέρασαν πέντε μήνες από το γεγονός στην Μάλτα και δυστυχώς η έρευνα, οι ερευνητές ε, έχουν ε, αρκεστεί με τα πορίσματα ότι η δολοφονία διαπράχθη από τη μαφία. Ποιος ε, έδωσε την αδιαγή όμως είναι το θέμα για την δολοφονία. Και δεν προχωράει η έρευνα. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, έχω μια ερώτηση. Πώς αισθάνεστε για τη Μάλτα. Ξέρουμε ότι δύο μέλη της κυβερνήσεως έχουν εκτεθεί στα Panama Papers και από τις εκθέσεις των αρμοδίων φορέων ε, στη Μάλτα και θεωρούνται διεφθαρμένοι και εξακολουθούν να στην κυβέρνηση αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό συμβάλλει σε αξιοπιστία. Δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης για τις έρευνες. Ντάλι, ο Επίτροπος, ε, ταπεινώθηκε από την έρευνα ε, της Όλαφ και του φορέα της Μάλτας επέστρεψε στη Μάλτα δεν έχει διωχθεί και έγινε και σύμβουλος του Πρωθυπουργού του άλλου, μάλλον, του άλλου κόμματος. Παράξενο. Δεν σας ανησυχεί. Όταν ακούγονται πολλές φήμες για ιδιωτικοποίηση νοσοκομείων, διάφορες εταιρείες ε, και λογαριασμούς στις παρθένους νήσους, της Βρετανίας, ε, πετρέλαιο, Αζερβαϊτζάν, πώληση θεωρήσεων κλπ άδειε διαμονής κλπ. Ηλεκτρονικά παιχνίδια, κρυπτονομίσματα κλπ. Όλα αυτά ε, είναι φήμε ότι όλα αυτά ισχύουν στη Μάλτα. Ποια είναι η απόψή σα από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτά που συμβαίνουν στη Μάλτα. Θέλω σαφήνεια για την ε, διάφορες τράπεζες, η τράπεζα, η τράπεζα Πιλάτους πήρε την άδεια παρά την ενδεχόμενη εμπλοκή σε υποθέσεις ξεπλήματος χρήματος από το Αζερβαϊτζάν αλλά και διασυνδέσεις με το Ιράν. Κλείνοντας, πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν είναι το σωστό μέρος για συζήτηση της διαφθοράς. Κανείς δεν διαρωτά τη διαφθορά σε αυτό το πλαίσιο, κυρίως το Κοινοβούλιο. Και το θέμα διασύνδεσης αυτού του θέματος με το κράτος δικαίου και με την εκταμείευση πόρων είναι πολύ σημαντικό. Και ναι, δεν θα ήμασταν εδώ τώρα, αν είχαμε δράσει για την Ουγγαρία εδώ και πολύ καιρό. Η Μπάρμπαρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους που είπαν ότι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι πιο θαραλέοι καθορίζοντας το κράτος δικαίου περί τίνος πρόκειται. Τι εννοούμε όταν μιλάμε για πολιτική διαφθορά. Γιατί πιστεύω κάτι τέτοιο. Όλοι γνωρίζουμε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι νομικοί, οι δικηγόροι, και ο νόμος υπηρετεί εκείνους που έχουν αναθέσει εκθέσεις εμπειρογνωμόνων. Και περιμένω τη λευκή βίβλος των δικηγόρων της Πολωνίας θα αποδείξει σαφώς ότι στην Πολωνία τα πάντα πηγαίνουν κατά γράμμα, σύμφωνα με το Σύνταγμα και ότι δεν υπάρχουν επιθέσεις κατά των δικαστών. Θα δούμε διάφορες αποχρώσεις της αλήθειας και της έλλειψης αλήθειας. Για να κατανοήσουμε τι γίνεται, θα πρέπει να εστιαστούν επί των υποθέσεων οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όχι η Επιτροπή της Βενετίας. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να εξασφαλίσουν το ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε την νομοθεσία μας επί των κοινών μας αξιών που αναφέρατε Επίτροπε. Και αν αυτή αποτελεί την αφετηρία μας, αν συμφωνούμε με αυτό, θεωρώ ότι η κατάσταση στην Πολωνία επουδενή δεν είναι καλύτερη από ό,τι ήταν την προηγούμενη φορά που την συζητήσαμε. Αν ο Πολωνός Πρωθυπουργό λέει ότι η Πολωνία ε, δεν είναι πλέον δημοκρατική χώρα που επικρατεί το κάτος δικαίου αλλά μιλάμε για δημοκρατικό εθνικό κράτος, αν το λέει αυτό ο Πρωθυπουργό, αυτό σημαίνει ότι αποκλίνουμε από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όπως τις αντιλαμβανόμασταν ε, παλιά. Και αυτή η ε, προσέγγιση ίσως να διαδοθεί και σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ο κίνδυνος και είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να εξασφαλίσουμε το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα εργαστούν δεόντως και ότι θα επεξεργαστούν τους ορισμούς περί κράτους δικαίου και περί διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής διαφθοράς. Ευχαριστώ. Λόπες Αγγιλάρο. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Επιτροπέ. Ξέρετε δεν μπορούμε να σας πούμε πόσοι από εμά υποστηρίζουν πραγματικά τα θέματα τα οποία αντιμετωπίσατε και τα οποία θίξατε στη σημερινή συνεδρίαση και πόσο πολύ πραγματικά σας υποστηρίζουμε και πόσο σας καλωσορίζουμε και εσάς και τις δράσεις σας για τα θέματα αυτά. Αλλά προκειμένου να είμαστε συμπληρωματικοί σε σχέση και με αυτά που ήδη ακούσαμε του συναδέλφου, να σα πούμε το εξή, ότι όλε αυτέ οι ανησυχίε και η Πολωνία, αλλά κυρίω η Πολωνία και η Μάλτα και η Σλοβακία μάλλον, αποτελούν, αν θέλετε, ένα σταυροδρόμι. Δεν συνδέονται όμω ε, το διευθυντικό θέμα στο χαρτοφυλάκιό σας που είναι η επιδείνωση του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ποιότητας της ίδιας της δημοκρατίας. που απειλούνται από την ε, επανελειμμένη και συρροή παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων. Άρα, εμείς δεν θέλουμε να δείξουμε μόνο τα θέματα αυτά θέλουμε να δείξουμε και την ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2018. Μήπως ανησυχείτε ότι είναι η τελευταία ή ίστατη ευκαιρία στη θετία της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου όπου μπορούμε να κάνουμε μια διαφορά. Όλη αυτή η νομοθεσία δηλαδή η οποία συστηματικά μπλοκάρεται από το Συμβούλιο Βίζες, Σέγγεν, όλα αυτά τα θέματα στην ατζέντα έχουν μπλοκαριστεί και δεν υπάρχουν πλέον πολλές ελπίδες να απελευθερωθεί ο δρόμος για την ε, δρομολόγησή τους. Και θα ήθελα λοιπόν να σκεφτείτε τι θα κάνετε και τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς για τα πολύ σημαντικά αυτά ζητήματα. Γιατί πολλοί από εμάς σας υποστηρίζουν σε ό,τι αφορά την Πολωνία. Ποιε είναι οι προοπτικές για την ε, συμπερίληψη του Κοινοβουλίου βάσει του 7-2. Γιατί το 7-1 δεν συμπεριλαμβάνει το Κοινοβούλιο. Το 7-2 όμω συμπεριλαμβάνει και η ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να αποφασίσετε μέχρι το τέλο τη θετίας κατά πόσον το Κοινοβούλιο όμω θα έχει δικαίωμα να ψηφίσει για τα θέματα αυτά. Κυρία Ρουίς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τίμερμαντς, Ξέρετε ότι σας εκτιμάμε όλους ιδιαίτερος εδώ. Ε, παράλληλα όμως μας φαίνονται πολύ ωραία γελικά πλασμένα όλα αυτά που μας είπατε όσον αφορά ε, το Λονδίνο, το, την δολοφονία που έγινε με ένα αέριο που είναι ρωσική παραγωγή. Οπότε ε, είναι ανέκδοτο. Προφανώς το κάναν όπως το κάναν η Βρετανική κυβέρνηση χρειάζεται την στήριξή μας ε, απόλυτα και έντονα. Δεύτερον, συγγνώμη, δεν θέλω να υπάρξει παρεξήγηση από αυτού, λέει ο κύριος Τίμερμανς. Εγώ είπα ξεκάθαρα ότι παρακολούθησα τη δήλωση της Τερέσα Μέη στην Βουλή των Κοινοτήτων και τη στηρίζω. Δεν έχω κανένα λόγο να διαφωνήσω με καμία λέξη από όσε πρόφερε. Οπότε μην υπάρχει παρεξήγηση από αυτού. Ακούσαμε ότι στηρίζεται τα όσα είπε η κυρία Τερέσα Μέη. Αλλά δεν φαίνεται έναν ατύχημα αυτό που έγινε, έτσι δεν είναι, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για ατύχημα. Και σας το λέω με κάθε συμπάθεια. Έχει σφραγίδα το γεγονός, θέλω να πω. Και συγγνώμη αν σας έφερα σε δύσκολη θέση. Τώρα. Είπαν οι συνάδελφοι και σας το είπα και εγώ πριν πόσο πολύ σας εκτιμάμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να ζητάει και απαιτεί έναν διάμεσο μηχανισμό ανάμεσα στο 7-2 και τη σημερινή κατάσταση. Γιατί βλέπετε ότι συσσωρεύονται οι περιπτώσεις και οι χώρες που τολμούν και πλήττουν θέματα πολύ βασικά για τη δημοκρατία στις χώρες μας. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητήσαμε λοιπόν μηχανισμούς, τους εγκρίναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν εφαρμόζονται. Αυτό είναι το ένα. Από την άλλη, κύριε Τίμερμανς, όταν διώκονται οι δικαστές, αυτό είναι εκφοβισμός και αυτή είναι η χειρότερη και πιο σοβαρή απειλή, όπως είπατε κι εσείς. Δεν θα υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις στα τέλη του μήνα, οπότε τι θα κάνουμε. Εγώ προέρχομαι από ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει υποστεί αυτόν τον εκφοβισμό. Βόρεια Ισπανία, στη χώρα των Βάσκων. Και επίσης υπήρχε δίωξη των δημοσιογράφων για να σιωπήσουν, τους δολοφονούσαν, Πρέπει να ξεφύγουμε από τους διαλόγους. Δεν φτάνουν. Όλο και περισσότερες χώρες προστίθενται στον κατάλογο. Σας το λέμε αυτό εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί σας στηρίζουμε. Θα συνεχίσουμε όμως να ζητάμε αυτά που ζητάμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριος Ράντα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε σας ευχαριστώ πολύ για την σαφή σας ε, στάση υποστηρίζοντας το κράτος δικαίου σε όλες τις χώρες μέλη. Πράγματι, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου αποτελούν τις βασικές αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι καθήκον όλων μας να τις προστατεύουμε, να τις σεβόμαστε, ε, να τις στηρίζουμε. Είτε είμαστε πολιτικοί, είτε απλός κόσμος. Βέβαια, φάνηκε πρόσφατα ότι δεν έχουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς για να προστατεύουμε τη δημοκρατία. Γι' αυτό και ζητάμε και φροντίσαμε να έχουμε αυτό το μηχανισμό τελευταία για την στήριξη του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Ελπίζαμε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο που μας πέρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είχε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν το έχουμε όμως. Μπορείτε λοιπόν να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες. Τι πρόοδος έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα από αυτού. Και μπορείτε να λάβετε υπόψη σας, σας παρακαλώ, και την επιμονή μας για αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία εφαρμόζονται εξίσου σε όλες τις χώρες μέλη, χωρίς πολιτικές προτιμήσεις υπέρ της μιας ή της άλλης χώρας. Και να σκεφτούμε και τον μηχανισμό για την Ρουμανία και την Βουλγαρία Ο έλεγχος της διαφθοράς, μήπως θα μπορούσε και αυτό να αντικατασταθεί από έναν τέτοιο μηχανισμό. Τέσσερα άτομα παραμένει παρακαλώ, να μείνετε κάτω από τα δύο λεπτά όμως, γιατί δεν θα ακούσουμε στη συνέχεια των, τις απαντήσεις του, του Επιτρόπου. Κύριε Ευχαριστώ Κλοντ, ευχαριστώ Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Στο πρόγραμμα εργασιών για το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλαμβάνει βασική έννοια το μέλλον τη Ευρώπη εξαρτάται από τη δυνατότητα να προσπιστεί τι κοινέ αξίε που μα ενώνουν. Δημοκρατία, το κράτο δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Περιμένουμε με ανυπομονησία και την εφαρμογή του κράτου δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι η ερώτησή μου είναι η εξή. Η πρότασή σα θα είναι φιλόδοξη όσο και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 2016 όσον αφορά το μηχανισμό για θέματα δημοκρατία κράτο δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα που εγκρίναμε μόλι τώρα. Ε, δεν θεωρείτε ότι μόνο μια ισχυρή στεναρή πρωτοβουλία θα επιτρέψει να εξισορροπήσει τους εγωισμούς και την αλαζονία κάποιων κρατών μελών και την παρέκκλησή τους και που, δεν, που αγνοούν και τις αποφάσεις του ΔΕΚ. Δεύτερη ερώτηση για τη μετανάστευση. Μπορούμε να προβλέψουμε το περιεχόμενο της δευτέρας εκθέσεως προόδου που σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο που θα αύριο. Τέλος, όσον αφορά τις διακρίσεις Έχουμε επανειλημμένε περιπτώσει ξενοφοβία, ρατσισμού και διακρίσεω που καταγράφονται σχεδόν καθημερινά σε όλα τα κράτη-μέλη. Δεν θεωρείτε, κύριε Επίτροπε, ότι θα χρειαζόταν πιο αποφασιστική δράση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε μια ερώτηση που συνέταξα εδώ και μερικέ εβδομάδε, ζήτησα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα πει αν θα μα παρουσιάσει μια στρατηγική για να αντιταχθεί ε, στην αφροφοβία, αφρικανοφοβία. Και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η προσωπική σα άποψη. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ λυπάμαι, που καλούμαστε να συζητήσουμε και πάλι για μία ακόμα φορά την Πολωνία. Αλλά πιστεύω, όπως είπατε, μπορούμε να προστατεύσουμε το, το κράτος δικαίου αν το κάνουμε ξεκάθαρα. Να μιλήσουμε λοιπόν ξεκάθαρα, όχι μόνο εκεί που απειλείται το κράτος δικαίου, αλλά και σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα. Χαίρομαι λοιπόν και είμαι ευγνώμων που όλοι συμμετέχετε και που τα συζητάμε όλα αυτά από κοινού, γιατί αυτή είναι η ένωσή μας και θα πρέπει να υπάρχουν κοινά πρότυπα για την ανεξαρτησία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το καθεξής. Το πρόβλημα είναι ότι όσοι εκφράζονται σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα αυτά στη χώρα μας ε, τους ε, καταδιώκουν, κατασκοπεί τους, ε, τους αποκαλούν κατασκόπους, τους απειλούν, ακόμα και με θάνατο, με δίωξη, τα ξέρετε αυτά ενδεχομένω. Και πρόκειται λοιπόν πραγματικά για παρενόχληση. Κάποιος ανέφερε την παρενόχληση των δικαστών, ιδιαίτερα αυτών που έρχονται στις Βρυξέλλες και άκουσα πρόσφατα ότι παρενοχλούνται και εκφοβίζονται οι γυναίκες τους, οι, γυναίκες, οι άνδρες τους, οι δημοσιογράφοι έχουν χάσει σχεδόν όλη τη δουλειά τους ε, σε περίπτωση που έχουν μιλήσει ανεξάρτητα. Όταν λοιπόν ε, Μίλατε για μια κρίση πολλών χωρών, γιατί κάποιος ε, ανέφερε μια λίστα χωρών. Ίσως ε, αυτό να αποτελεί μια δραματική παρουσίαση του πόσο ευάλωτη είναι αυτή η ελευθερία τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Σε όλες τις χώρες αυτές η συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας τελικά επιζητά δημοκρατία, επιζητά αυτά τα δημοκρατικά πρότυπα και χαίρομαι που με την Επιτροπή αυτή υποστηρίζονται τα εργαλεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία έχουμε ήδη συζητήσει. Αυτό πραγματικά μπορεί να ενισχύσει την ε, κοινωνία των πολιτών και ελπίζω πραγματικά να ενισχυθούν έτσι όλα τα εργαλεία αυτά που χρειάζονται. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κώστερ, αλλά για δύο λεπτά και όχι παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Επιτροπέ, δύο σημεία ήθελα να αναφέρω. Καταρχάς την κατάσταση στην Πολωνία και την Ουγγαρία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ δραστηριοποιείται δραστηριοποιείται για την ανεξαρτησία των δικαστηρίων, για την ε, διάκριση των εξουσιών και θα πρέπει λοιπόν να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ε, γίνεται στην Ουγγαρία και στην Πολωνία να εκλέγονται από πολλούς πολίτες κόμματα τα οποία σχηματίζουν κυβέρνηση και τελικά υποσκάπτουν αυτό το κράτος δικαίου. Έχει να κάνει αυτό με την πολιτική λιτότητα του παρελθόντος από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την ευρωπαϊκή πολιτική, το γεγονός ότι ο κόσμος ε, αποστρέφεται τελικά τη δημοκρατία και εκλέγει κόμματα για τα οποία δεν παίζει μεγάλο ρόλο η δημοκρατία. Τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι θα έπρεπε να κάνει προκειμένου να ανισχυθεί η δημοκρατία στην Πολωνία, να ανισχυθούν και αυτοί που γίνουν στους δρόμους και διαδηλώνουν στην Πολωνία δηλαδή για την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Δεύτερο θέμα. Δείξτε το θέμα της διαφθοράς, του ξεπλήματος χρήματος. Χρήματα από διαφθοράς και από νομιμοποίηση παράνομων ε, προσόδων. Το θέμα των πληροφοριοδοτών που αποκαλύπτουν τέτοιες περιπτώσεις. Τι έχει γίνει για την προστασία αυτών. Είχαμε κάποιες προτάσεις πέρσι. Τι έγινε με αυτές τις ε, συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάζα τελευταίος. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Αντιπρόεδρε Τίμερμανς, ε, και εσεί και άλλοι συνάδελφοι μας υπενθυμίσατε ότι τους τελευταίους έξι μήνε δολοφονήθηκαν, εκτελέστηκαν δύο δημοσιογράφοι σε μία απόπειρα να τους βάλουν φήμουτρο για τι εργασίε του, για την έρευνά τους, για τη διαφθορά στις δύο χώρες και άλλοι έχουν απειληθεί και οι επιχειρήσεις ε, Παίρνουν σε τεράστια έξοδα για να εκφοβήσουν ε, ενδεχόμενους ε, ε, πληροφοριοδότες με τεράστια δικαστικά έξοδα. Αυτό συμβαίνει, συνέβησαν και στην περίπτωση της Μαλτέζας δημοσιογράφου και σε άλλες περιπτώσεις. Και έτσι Αντιπρόεδρε Τίμερμαν, σας κάλεσαν να προτείνετε μία οδηγία για την προστασία των δημοσιογράφων προτείνετε, θα σκοπεύετε να προτείνετε λοιπόν μια τέτοια α, οδηγία και αν όχι, τι μέτρα μπορεί να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προστατεύσει από τέτοια μέτρα τους α, ε, δημοσιογράφους και τι δουλειά έχει κάνει η Επιτροπή με την έκθεση για τη Μάλτα και το κράτος δικαίωση Μάλτα στις 31 Μαρτίου του χρόνου αυτού και ευχαριστώ και να σας πω ότι αυτή την ε, εβδομάδα κύριε Επίτροπε θα γίνει η συζήτηση για τη Σλοβακία. Να θα θέσω λοιπόν ένα πολύ γρήγορο ερώτημα. Όταν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση και αυτό συνέβη στη Σλοβακία, σε τελική ανάλυση ελπίζουμε να δούμε κατά πόσον υπήρξε ανάμειξη του κράτους αν θα υπάρξει συγκεκριμένη υπόδειξη αυτού, αλλά πάντα θα υπάρχει η υπόνοια αυτή και θα επικρατεί και έλλειψη εμπιστοσύνη. Ποια είναι η αποψή σα λοιπόν ω τώρα. Νομοθεσία για τους δημοσιογράφους, για προστασία ή μόνο να κοιτάξουμε την διάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πώς θα προστατεύσουμε λοιπόν τους, ανθρώπου, πώς αντιμετωπίσουν αυτά τα θεμελιώδη προβλήματα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την εμπιστοσύνη στην προστασία των δημοσιογράφων. Αυτό ισχύει και για τη Σλοβακία και για εσά. Θα θέλαμε να ξέρουμε και την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α αρχίσω με αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλού από εσά. Όταν ε, αρχίσαμε να κοιτάμε αν μπορούμε να προτείνουμε νέα νομοθεσία, προσοχή, πρέπει να δούμε τι αρμοδιότητες έχουμε ε, σε αυτό το πεδίο. Γιατί μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις από τις χώρες μέλη. Το μελετάμε αυτό. Αλλά Κλόντ είναι δύσκολη ερώτηση για να την απαντήσω έτσι τώρα αμέσω. Υπάρχει το θέμα της προστασίας των δημοσιογράφων και θα επανέλθω σε αυτό βέβαια, αλλά υπάρχει και το θέμα της χρήσης όλων των εργαλείων, των μέσων που διαθέτουμε ήδη, ώστε όταν κάποιος ερευνά μια υπόθεση, να μην διώκει τους ε, υπεύθυνου ή την διαφθορά ή τις συνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσα διαθέτουμε, ώστε αυτά να τα κάνουν η Eurojust, η Europol, το Συμβούλιο της Ευρώπης. Εγώ δεν βλέπω κανένα πρόβλημα στη συνεργασία θεσμικών οργάνων και μηχανισμών που έχει φτιάξει το ε, Συμβούλιο της Ευρώπης να συνεργαστούμε με τους άλλους. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε όμως μας να το κάνουμε, αλλά δεν βλέπω να είναι κακό να πρέπει να κάνουμε κάτι που έχει ήδη γίνει, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πρέπει να κάνει κάτι που έχουν ήδη κάνει οι ειδικοί στην Επιτροπή της Βενετίας, που είναι αξιοσέβαστη παντού, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό που ρωτάτε είναι τόσο θεμελιώδες, που δεν μπορώ να πω ότι έχω μια έτοιμη απάντηση σήμερα. Αλλά πρέπει να καθίσουμε και να σκεφτούμε πώς θα οργανώσουμε καλύτερα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, ώστε να μπορούμε πιο εύκολα να τα χρησιμοποιούμε. Δεν υπάρχει καμία χώρα που να μην έχει ζητήματα με το οργανωμένο έγκλημα ή με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Είτε πρόκειται για τον πολιτικό έλεγχο, τον οικονομικό οτιδήποτε. Παντού μπορεί να υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Οπότε, όταν ετοιμάσουμε το έγγραφό μα για τα τέλη τη χρονιά όσον αφορά την πλαισίωση του νόμου δικαίου, του κράτου δικαίου, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά που έχετε πει και εσεί στο ψήφισμά σα για το πώ μπορούμε να γενικεύσουμε αυτά τα θέματα. Άρα δεν πρόκειται για τις χώρες μέλη μόνο για τις οποίες μιλήσαμε σήμερα, πρόκειται για ένα πιο οριζόντιο θέμα που έχει να κάνει με όλες τις χώρες μέλη και η εξουσία μας θα ενισχυθεί αν έχουμε ένα μέσο που να μπορούμε οριζόντια να χρησιμοποιήσουμε σε όλες τις χώρες μέλη. Οπότε δεν θα είναι το αν έτσι, αν αλλιώ αν αλλιώτικα. Αν είναι πιο οριζόντιο το μέσο που θα διαθέτουμε, πιστεύω ότι θα ενισχύσουμε τα επιχειρήματά μας. Δεν υπάρχει καμία χώρα μέλος που να είναι υπεράνω μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες έχουν τέτοια ζητήματα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή είπαμε Μάλτα, Σλοβακία, εμείς ζητάμε μια κοινή ερευνητική ομάδα με την Europol. Για τελειώς πώς θα καλύψετε όλα τα θέματα διαφορετικά και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο. Και εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, να ξέρετε. Ωραία. Και για να είμαι και ε, δίκαιος και για τις δύο αυτές χώρες, και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν διεθνή στήριξη. Μερικές φορές τη ζήτησαν, άλλες φορές την ε, έλαβαν απευθείας και το θέλανε και δύο. Καμία δεν είπε, όχι αυτό είναι δικό μας εθνικό ζήτημα και δεν θέλουμε να ανακατευθείτε. Όχι, δέχτηκαν ε, τη διεθνή βοήθεια είτε από τη Scotland Yard, είτε από την Eurojust, την Europol. Και αυτό είναι ο σωστό τρόπο, γιατί μόνο έτσι γινόμαστε πιο δυνατοί. Ξέρουμε ότι το οργανωμένο έγκλημα καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά το ωφέλη της εσωτερικής αγοράς. Το οργανωμένο έγκλημα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο καλύτερος φορέας στην ε, εσωτερική αγορά αν δεν φροντίσουμε αυτοί που καταπολεμούν το ε, διεθνές έγκλημα να καταλάβουν πώς λειτουργεί η εσωτερική αγορά, θα χάσουμε τον αγώνα. Και δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Πρέπει οι αρχές που διώκουν το έγκλημα να συνεργάζονται μεταξύ τους και να υπάρχει και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Γιατί δεν έχουν πάντα εμπιστοσύνη για ανταλλαγή πρακτικών, για συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό έχει άμεση σχέση με το κράτος δικαίου. Και έρχομαι και στα μέσα ενημέρωση τώρα γενικότερα. Όπως είπατε και συζητήσαμε, πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν αρχίσαμε αυτό το ωραίο ταξίδι, εγώ τη δεκαετία του 80 που θυμάμαι βγήκα από το πανεπιστήμιο και κάποιος φοιτητής, η φοιτήτρια μάλλον, είπε ότι θα επανενωθεί η Γερμανία και γελάσαμε. Ε, μα ε, αρέσει τόσο πολύ η Γερμανία που πολύ χαιρόμαστε που έχουμε δύο. Ποτέ ήταν αδιανόητο για μα να ενωπηθεί η Γερμανία και όμω έγινε. Δείτε λοιπόν αυτό το υπέροχο ταξίδι που κάναμε. Τώρα λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πρόκειται για μια γραμμική πορεία με μία κατεύθυνση. Δεν είναι δεδομένο ότι πάντα θα πηγαίνουμε μπροστά. Και δεδομένη τη κρίση την οποία περάσαμε, την οικονομική, την τραπεζική, τη μεταναστευτική, η τρομοκρατία, αντιδράσεις του κόσμου. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν και σε άλλα, στην αμφισβήτηση της ίδιας της δημοκρατίας. Η δημοκρατία με εξυπηρετεί, όχι. Υπάρχουν εναλλακτικέ. Οπότε δεν φτάνει να μένει ο καθένας με το δικό του υπόβαθρο. Το βλέπω και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι κάποιοι θαυμάζουν τον Πούτιν. Μα πώς είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει εκεί, να αρχίσουμε να θαυμάζουμε κάποιον που ακολουθεί τέτοιες πρακτικές. Και όμως συμβαίνει και εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως το ξέρουμε. Και πρέπει να συμφωνήσω με τον κύριο Κώστορ εδώ ότι υπάρχει ένα πιο βασικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχει να κάνει με τη λιτότητα. Έχει να κάνει σίγουρα με την κρίση, ναι. Έχει να κάνει με αυτούς που έχουν στραμμένη την πλάτη στο μέλλον γιατί νιώθουν ότι δεν έχουν μέλλον και προσελκύονται από κάποιους που τους εμφανίζουν ένα παρελθόν που είναι καλύτερο από οτιδήποτε άλλο και έτσι φτάνουν στον εθνικισμό και όταν φτάνουμε στον εθνικισμό έχουμε την ξενοφοβία, βλέπουμε τον αντισημιτισμό, βλέπουμε τόσο κόσμο να νιώθει ότι ο άλλος είναι απειλή για αυτόν. Και αυτό είναι που διακυδεύεται σήμερα. Είναι κάτι παραπάνω από μεμονωμένες περιπτώσεις. ευχαριστώ να τις συζητήσω. ήθελα να σας εξηγήσω Πώς βλέπω εγώ το ζήτημα ότι είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Σε πολλές χώρες υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Οι πολιτικοί αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης ε, αρνητικά, ως απειλή. Μήπως με κάνουν ε, να χάσω τις επόμενες εκλογές. Τι να κάνω, να τους εκφοβήσω, να τους σιωπήσω, να χρησιμοποιήσω μέσα ώστε να μην μιλήσουν ποτέ με άσχημο τρόπο για μένα. Και χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα. Και έχουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που βέβαια δεν ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. Και χαίρομαι για την έκθεση που έχουμε σήμερα στα χέρια μας με κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να συμπεριφερθούμε απέναντι στα μέσα κοινωνικής ε, δικτύωσης. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο των fake news. Χωρίς ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης δεν μπορούμε να έχουμε δημοκρατία. Μπορείτε να έχετε μια μορφή δημοκρατούρ, όπως στη Ρωσία, που πάτε, ψηφίζετε και δίνετε την εντύπωση ότι ζείτε σε δημοκρατία, αλλά δεν υπάρχει αντίβαρο. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε στους αυτούς μας να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Είναι πολύ βασικό να σεβόμαστε αυτούς που χάνουν τις εκλογές αυτού που δραστηριοποιούνται σε άλλους κλάδους. Ο πολιτικός σας αντίπαλος είναι αντίπαλος, δεν είναι εχθρός. Αυτή λοιπόν την πολιτική νοτροπία, το να δεχόμαστε να διαφωνήσουμε με τον άλλον, έχουμε αρχίσει να την ξεχνάμε. Σε μερικέ χώρε μέλη πολύ εύκολα θεωρεί κανεί εχθρό του κράτου όποιον είναι πολιτικό του αντίπαλο. Αυτό όμω δηλητηριάζει τη δημοκρατία γιατί τότε τον πολιτικό σας αντίπαλο το βγάζετε από το σύστημα. Και αυτό είναι το τέλος της δημοκρατίας. Γιατί είναι δηλητηριώδες αυτό, γιατί αυτό σημαίνει ότι εσείς ε, νιώθετε τόσο μεγάλη την απειλή του να βρεθείτε εσείς εκτός του πολιτικού συστήματος, να χάσετε τις εκλογές δηλαδή, που σας κάνει να συμπεριφέρεστε παράλογα. Ωραία. Πέντε-έξι εκλογές Κάποιο χάνει τις εκλογές. Μα χρειάζεται μια ισχυρή αντιπολίτευση, όπως χρειάζεται και μια ισχυρή κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, δεν έχετε καν ισχυρή κυβέρνηση. Και σε αυτόν που αναφέρθηκε στις κάτω όσοι δρούν εκτός του νόμου, διώκεται από τον νόμο στις κάτω και για να απαντήσω στον κύριο Γιούρεκ, αν έπρεπε να θέσω τώρα το θέμα της άμβλωσης στην Πολωνία, τι θα μου λέγατε, α μην ανακατεύεστε, δεν είναι δικό σας θέμα. Και σε έναν βαθμό θα είχατε δίκιο. Οι εθνικές αρμοδιότητες είναι εθνικές αρμοδιότητες και πρέπει να το σεβαστούμε. Και εγώ προσωπικά τώρα το κάνω εγώ το σχόλιο, οι Πολωνές πρέπει να προσπαθήσουν να πετύχουν αυτό που θέλουν στην Πολωνία, εντάξει. Αλλά αν υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτά πρέπει να προχωρήσουμε. Το θέμα της αυθανασίας δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπα και πριν στις κάτω χώρες, αν κάποιος παραβιάσει τον νόμο θα διωχθεί. Το λέω γιατί γνωρίζω πολύ καλά την περίπτωση των κάτω χωρών. για τους κανόνες του προπολογισμού και αν πρέπει να υπάρχει αιρεσιμότητα, υπό προϋποθέσεις δηλαδή. Ειλικρινά πιστεύω ότι αν υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά το κράτος δικαίου, θα πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίες και για το κατά πόσο δαπανώνται σωστά τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα διαρθρωτικά ταμεία, έχει να κάνει με όλες τις πληρωμές που κάνουμε, με χρήματα τα οποία συγκεντρώνονται από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Άμεσες ενισχύσεις, άλλες πληρωμές διασυνοριακά. Επίσης ξέρω ότι είναι δύσκολο και περίπλοκο να το διατυπώσει αυτό νομικά, γιατί πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα, να αντιμετωπίσεις δηλαδή αναλογικά το πρόβλημα που προσπαθείς να αντιμετωπίσεις. Οπότε εγώ δεν το βλέπω αυτό σαν ένα κυπροκό, δηλαδή αν δείξεις αλληλεγγύη εκεί δεν θα πάρεις χρήματα αλλού. Όχι, δεν λέω ότι έτσι πρέπει να προχωρήσει το σύστημα. Βλέπω όμως τη δυνατότητα που χρειάζεται μελέτη να έχουμε σαν γενική αρχή τον κανόνα που λέει ότι αν δεν είμαστε σίγουροι ότι τα χρήματα δαπανώνται βάσει κανόνων, δεν πρέπει να δαπανώνται. Και ειλικρινά πιστεύω, θα ήθελα να ενθαρρύνω όλες τις χώρες μέλη να συμμετάσχουν στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής εισαγγελία. γιατί μπορεί να εξετάσει κατά πόσο δαπανώνται σωστά τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Φορολογούμενου, όπαξ και υπάρχουν αμφιβολίες. Πολύ σημαντικό λοιπόν. Και μπορείτε και τον αντιστρέψετε, λέω, σαν ιδέα. Αν δεν θέλετε να συνεργαστείτε με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, ε, τότε για να δούμε. Πρέπει να μπορείτε να συμμετέχετε στο δημοσιονομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δηλαδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν δαπανάτε τα χρήματα σωστά. Και επανέρχομαι στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οι εθνικοί δικαστές είναι Ευρωπαίοι δικαστές στον τρόπο με τον οποίο ασκούν το επαγγελμά του. Αν δεν ξέρουμε λοιπόν κατά πόσο είναι ανεξάρτητοι αυτοί οι δικαστές ή ότι κατά πόσο αυτό που κάνουν έρχεται μετά από εντολή της κυβέρνησής τους, ε, πώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μπορεί να διασφαλίσει ότι με ανεξαρτησία οι εθνικοί δικαστές κρίνουν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν ο εθνικός δικαστής που είναι και ευρωπαίος δικαστής να μπορεί να ε, προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο χωρίς να παρεμβαίνει κανένας κυβερνητικός φορέας. Γι' αυτό είναι πολύ καλό που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου έβγαλε την απόφαση αυτή που αυτό το αποσαφηνίζει. Το ζήτημα τώρα που τέθηκε, ένα ακόμα ζήτημα, είναι το θέμα των ε, δράσεών μας απέναντι στην Ουγγαρία. Δεν αναφέρθηκα πριν στην Ουγγαρία, την προηγούμενη φορά το έκανα. Να το ξαναπώ. Είμαστε κατά της Ουγγαρίας για θέματα που έχουν να κάνουν με την νομοθεσία ε, για την ανώτατη εκπαίδευση, για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, για το άσυλο και άλλα. Θα συνεχίσουμε. Δεν θέλω να έχετε αμφιβολίες από αυτού. Το κάνουμε. Και θα συνεχίσουμε. Αλλά και εδώ θέλω να κάνω μία παρατήρηση για την πολιτική νοοτροπία. Δεν παίρνουν όλα ε, στη δικαστική διένεξη δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μιλάτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ε, πώς μιλάτε για ανθρώπους διαφορετικής φυλής. Όλα αυτά επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος δικαίου στη χώρα σας. Επηρεάζει τη δημοκρατική κοινωνία. Και εδώ πιστεύω ότι ακριβώς γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση με την Ουγγρική κυβέρνηση και τις Ουγγρικές αρχές. Προσβλέπουμε επίσης να δούμε κατά πόσο αυτή η νομοθεσία της όρος είναι συμβατή ή όχι. Θέλουμε να το διευκρινίσουμε και αυτό. Το ερώτημα της κυρίας Έρνης, κατά πόσο οι συνθήκες, οι συνθήκες ακόμα επαρκούν. Νομίζω ότι απάντησα, δεδομένη και της ευρύτερη εικόνα που έδωσα προηγουμένως στην απάντησή μου. Οι συνθήκες, ξέρετε, είναι σαν να παίζουν ένα μάτσα. Αν οι ποδοσφαιριστές αποφασίσουν όλοι μαζί να αγνοήσουν το διευθυντή, τι νόημα έχει, έχουν οι κανόνες. Είναι τμήμα της δημοκρατικής κουλτούρας, της κουλτούρας του κράτους δικαίου στην Ευρώπη ότι σεβόμαστε τις συνθήκες τις οποίες έχουμε προσυπογράψει. Αν ε, όχι, τα δικαστήρια που φαίνονται αναλόγως και θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις και δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα θυσιάζουμε όλα αυτά στο βόμο της εθνικής επικυριαρχίας. Εδώ θα πρέπει να δείξουμε προσοχή γιατί όταν κανείς δεν σέβεται το κράτος δικαίου ε, παραβιάζει και πολλά άλλα πράγματα, όχι μόνο ένα-δύο κανόνες, αλλά την ίδια τη δομή, την φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit και τη διατήρηση του χάρτη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των θεμελιδών δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, είτε είναι Βρετανοί είτε όχι. Είναι λυπηρό και τραγικό αυτό το Brexit. Πόσο μάλλον αν οδηγήσει και στην επιδείνωση των δικαιωμάτων των πολιτών όπως υφίστανται σήμερα η τραγωδία θα ήταν ε, έτσι περαιτέρω μεγαλύτερη. Θα πρέπει λοιπόν να αντιτηρηθεί η προστασία του χάρτη των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η κυρία Άντερσον ε, επεσήμανε κάποιες ε, αναφορές στα έγγραφα. Θα τις εξετάσουμε για να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κυρία Κόμμα έκανε πολύ συγκεκριμένε ερωτήσει για πολύ συγκεκριμένα θέματα στη Μάλτα. Δεν έχω τόσο συγκεκριμένε πληροφορίε, τόσο συγκεκριμένα δεδομένα να σα απαντήσω για τα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που κάνατε. Υπάρχει σχετική έκθεση, αναφορά και σας εγγυώμαι ότι θα συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε, να συζητάμε με την ε, Μαλτέζικη κυβέρνηση ο Πρωθυπουργό όταν παρευρέθηκε σε μία σύνοδο γιατί ήταν 27 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που συμμετείχαν. Μίλησε και με τον Υπουργό, Εξωτερικών, τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και διαρκώς προωθώ τα θέματα αυτά και τους καλώ να συνεργάζονται για την ε, Λευκή Βίβλο τώρα, να πω δύο λόγια. Η Λευκή Βίβλος. Δημοσιεύτηκε με την τοποθέτηση της πολωνικής κυβέρνησης μας απεστάλλει και σε εμά και στο κοινό και σε όλα τα κρατημέλη. Θα ήθελα όποιος γνωρίζει, όποια οργάνωση γνωρίζει κατά παραπάνω, κάτι παραπάνω, να μας στείλει την άποψή του, το όραμά του, για να δούμε ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου. Και έλαβα απάντηση από κάποια κράτη-μέλη που μας είπαν ότι κοιτάξτε, μας αναφέρετε στη Λευκή Βίβλο, αλλά εξηγήστε παρακαλώ ποια είναι η δική μας τοποθέτηση. Αυτό είναι θετικό. Νομίζω ότι εμπλουτίζει τη συζήτηση προκειμένου να ενημερώνεται και ο κόσμος και η Λευκή Βίβλος αλλά και η ανταπόκριση, το πώς έγινε δεκτή η Λευκή Βίβλος από τα άλλα κράτη-μέλη. Και ελπίζω να διορθώσουμε τις ε, απόψεις που επικρατούν και ελπίζω, θα συνεχίσω μάλλον τη συνεργασία με τι πολωνικέ αρχέ. Αναμένουμε μεγαλύτερη διευκρίνηση από πλευρά τη πολωνική κυβέρνηση και ελπίζω να το επιλύσουμε τελικά το θέμα αυτό. Και δεν λέω κάτι καινούργιο προφανώ προ του Πολωνού ε, βουλευτέ ε, εδώ στην Επιτροπή. Γιατί στην τελική ανάλυση ο μοναδικό που μπορεί να το λύσει το θέμα είναι οι ίδιοι οι Πολωνοί. Εμεί να βοηθήσουμε, να δείξουμε τα όρια στα οποία μπορεί να φτάσει η πολωνική κυβέρνηση θα πρέπει να σεβαστεί το κράτος δικαίου, θα πρέπει να σεβαστεί ε, τα συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά στην τελική ανάλυση η Πολωνία, ο πολωνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα καθορίσει το μέλλον τους, είτε θα είναι ίδιο με κάποιες άλλους λαούς, είτε κατά πόσον θα διαφέρει. Εγώ ελπίζω από το βάθος της καρδιάς μου γιατί είναι ιδιαίτερη η περίπτωση της Πολωνίας, να ακολουθήσει η Πολωνία ε, το ευρωπαϊκό αυτό μονοπάτι. Δεν μπορώ να φανταστώ μια ασφαλή Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, αν προκληθεί μεγαλύτερος διχασμός μεταξύ μας. Ελπίζω λοιπόν αυτός ο διάλογος να οδηγήσει σε αποτελέσματα. Τελευταίο θέμα λοιπόν για τους πληροφοριοδότες. Ε, θέλουμε να καταθέσουμε σύντομα μία πρόταση και έχω ανοιχτή συζήτηση με διάφορους συναδέλφους μου λαμβάνουμε υπόψη τις απόψεις που εκφράστηκαν και στο Κοινοβούλιο και από άλλους ε, εμπλεκόμενους φορείς και από το Συμβούλιο της Ευρώπης και θα πρέπει να εξετάσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία, τις καταφυντήριες γραμμές, να δούμε τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση βάσει αυτών. Αναφέρθηκα στο θέμα της ξενοφοβίας, ε, του ρατσισμού που είναι σε άνοδο. Νομίζω ότι αν θέλουμε να δείξουμε ότι έχουμε μια απάντηση στο θέμα, το μεταναστευτικό, το προσφυγικό, το θέμα αυτό, ξέρετε, δεν πρόκειται να φύγει από μόνο του. Θα συνεχίσει η μετανάστευση για μια-δυο γενιές στην Ευρώπη. Και αν η απάντηση δική μας είναι να δημιουργήσουμε μια ήπειρο των παραμυθιών, όπου πιστεύουμε ότι με τύχη και με φράχτε θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα, νομίζω ότι το μέλλον τη Ευρώπη θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Θα στραφεί ο Ευρωπαίο κατά του Ευρωπαίου. Οι γείτονε θα ζητούν ελεημοσύνη. Θα φύγουμε από την λογική του win-win της ε, διπλής ωφέλειας και θα πάμε σε μια λογική Τραμπ εγώ κερδίζω και εσύ χάνει. Και μετά από δύο αυτοκτονικούς πολέμου, νομίζω ότι διδαχτήκαμε ότι η ευημερία μπορούμε να βρούμε μόνο μαζί. Αν όλα πάνε καλά, αν ε, αποταχθούμε την ιδέα αυτή και αν δημιουργήσουμε μια κατάσταση όπου θα θεωρούμε ότι το δικό μου έθνος μπορεί να ευημερήσει μόνο αν αποτύχει το δικό σου, αν πιστεύουμε ότι τελικά έχει δίκιο ο Πούτιν που παίρνει το χάος στις γειτονικέ του χώρε, αν αυτή την προσέγγιση επιλέξουμε στην Ευρώπη, ας ξεχάσουμε το κράτος δικαίου, αλλά ας ξεχάσουμε και την ευημερία και ας ξεχάσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το θέμα της μετανάστευσης είναι κρίσιμο. Αν εγκαταλείψουμε την ιδέα ότι αυτό το μπορούμε να το επιλύσουμε μόνο από κοινού ως Ευρωπαίοι και πιστέψουμε ότι αρκούν οι φράχτες, θα αποτύχουμε όλοι μαζί. Αυτή είναι η δική μου λοιπόν ιδέα για την ευρωπαϊκή συνεργασία, για τον εξυγχρονισμό των διατάξεων του Διβλίνου, για να υπάρχει καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα χάσουμε και την επαφή μας με την ανθρωπιά μας και να καταπνίξουμε την ανάπτυξη της ξενοφοβίας και του ρατσισμού στην Ευρώπη. Σας ζητώ συγγνώμη που με ακρηγόρησα. είπατε σας ευχαριστούμε. Uh, Ευχαριστώ συνάδελφοι για την ευγλωτία σας και τη συντομία σας. Με λίγη υπομονή θα ξεπετάξουμε και το επόμενο σημείο. Συμφωνούν συντονιστέ τον πίνακα για το σχέδιο ψηφίσματο εκ μέρου τη Επιτροπή στην Ολομέλεια. Θέμα οργανώσει κοινωνία των πολιτών στα κράτη-μέσα Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Αν έχετε χρόνο, πολύ γρήγορα μπορούμε αυτό λοιπόν το θέμα του ψηφίσματος να το εξετάσουμε. Στις 9 Απριλίου θα γίνει ψηφορία στη Λίμπε. Θέλουμε να εργαστούν γρήγορα οι ομάδες. Θέλει κάποιος να σχολιάσει. Μάικλ Μπόνι. Uh, that... Uh, Ευχαριστώ, Κλοντ. Άριστη συνέχεια της πρώτης συζήτησης, ο αντιπρόεδρος Τίμερμανς είπε ότι όλα εξαρτώνται στο κάτω-κάτω από τη στάση μας, στις χώρες μας. Εξαρτώνται από το πώς χρησιμοποιούμε τη δημοκρατία, πώς την υπερασπιζόμαστε, πώς πρασπίζουμε το κράτος δικαίου, πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε με θεμέλια τις αξίες. Έχουμε συζητήσει σε διάφορες ομάδες το θέμα αυτό και το ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Πώς θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της δημοκρατίας, της συμμετοχικής δημοκρατίας, πώς μπορούν να υπερασπιστούν τις αξίες μας. Και μετά την παρουσίαση της Υπηρεσίας για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, Διεφάνει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και έχουμε ένα συρρυκνούμενο χώρο για τις κοινωνίες των πολιτών στην Ευρώπη. Αναλύοντας όλα αυτά τα θέματα και συμμετέχοντας σε πολλές ε, συζητήσεις, δημιουργήθηκε η ιδέα συντάξεως ψηφίσματος. Γιατί είναι σημαντικό το ψηφίσμα. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε απάντηση. Να στηρίξουμε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να δημιουργήσουν το υπόβαθρο για δημοκρατία, για κράτος δικαίου και ασυμμετοχή των πολιτών στον πολιτικό βίο και στη δημόσια ζωή. Υπάρχουν κάποια εργαλεία. Λόγω όμως της αξιολογήσεως πολλών θεσμικών φορέων και της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομικής πολιτικής, βλέπουμε ότι τα εργαλεία αυτά δεν αρκούν. Χρειάζεται ειδικό εργαλείο αποκαλείται Ευρωπαϊκό Εργαλείο Αξίες Αξιών. Θέλουμε να συζητήσουμε τώρα αυτό το μέσο, διότι ταυτοχρόνως συζητούμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στην έκθεση που υπευλήθη από την Επιτροπή Προπολογισμών, κάποιοι από διάφορες πολιτικές ομάδες παρουσίασαν τροπολογίες Στο άρθρο 85α έχουμε μία σύσταση. Να... Στο έγγραφο έχει τίτλο Ευρωπαϊκό Ταμείο Δημοκρατίας στην Ενίσχυση και Υποστήριξη Κοινωνίας των Πολιτών και φορέων που εργάζονται στον τομέα της δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα χειρίζεται το Ταμείο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό είναι το δεύτερο σημείο μου. Σημαντικότατο το άμεσο εργαλείο και χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια, πρέπει να συζητήσουμε πολλά οικονομικά ζητήματα. Θα ήταν όμως πολύ καλό να έχουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Εργαλείο Αξιών που θα το χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημαντικότατο λοιπόν όταν συζητούμε τις οργανώσεις των κοινωνιών των πολιτών κυρίως στο τοπικό επίπεδο ε, να λάβουμε υπόψη ότι χρειάζονται στεναρή υποστήριξη. Σε πολλές ομάδες το συζητήσαμε το θέμα. Σημαντικότατο θέμα για όλους μας. Με αυτό το ψήφισμα και με την ακολουθούσα συζήτηση στην Ολομέλεια θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε στις συζητήσεις περί του μελλοντικού πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και μπορούν πραγματικά να στηρίξουμε το τρόπο τη οργανώση κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη. Ήσασταν όλοι πολύ υπομονετικοί. Δευτέρα, Στρασβούργο, τον αναγνωρίζω, θέλω να πάρετε τη συζήτηση. Έγινε τεχνική συζήτηση την Παρασκευή μετά την απόφαση των ιστών να προχωρήσουμε. Βέβαια, ο μηχανισμός αξιών και κλπ. είναι θέμα ευαίσθητο. Περιμένω οι ομάδες να το συζητήσουν εξαντλητικά και ταχαίως διότι έχουμε την 9η Απριλίου ως προθεσμία. Σύντομο χρονικό διάστημα για, την, ε, το ψήφισμα. Κύριε Στίβενς, έχετε κάτι να πείτε σε αυτό και Μπίρκιτ. Σύντομα παρακαλώ, σύντομα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να αντιδράσω στην πρόταση του κυρίου Μπόνι. Η δικιά μου αντιπροσωπεία, το ΕΝΒΕΑ, λέει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η τήρηση των βασικών αρχών. Αλλά έχει δεύτερε σκέψει για αυτή την πρόταση. Πρώτα απ' όλα γιατί οι μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις που προτείνουν αυτή την πρόταση υπονοούν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη δημοκρατία στην ε, Ευρώπη επειδή κάποιοι ψηφοφόροι κάνουν άλλε επιλογέ. Επιλογέ ε, όμω που δεν ικανοποιούν κάποιε μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Δεν είναι όμως δημοκρατικό το να μην μπορούν να εκφραστούν δημόσια όλες οι απόψεις χωρίς να επηρεάζονται. Και αυτό λοιπόν η πρόταση αυτή πιστεύω ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε κυβερνητικές απόψεις που θέλουν να προωθήσουν κάποιες ιδέες όπως στην Τουρκία και στην Ισπανία. Αναρωτιέμαι κατά πόσο είναι αυτό σωστό ή επιβάλλει κάποια ορθή πολιτική σκέψη μόνο. Συμφωνώ ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η ξενοφοβία, αλλά θα πρέπει να είναι δυνατό να καταλήξουμε κάπως όσον αφορά την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη. Το ότι υπάρχουν κόμματα ευρωσκεπτικιστικά σε διάφορες χώρες δεν σημαίνει ότι υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας. Αντίθετα σημαίνει ότι η, δημοκρατία δεν, η, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρνει να προσφέρει στους πολίτες αυτό που θέλουν, που είναι ελευθερία, απασχόληση και αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια δημοκρατία που να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των πολιτών και αν αυτό γίνει δεν χρειάζεται αυτό που προτείνει ο κύριος Μπόνη. Θέλω λοιπόν να μην βιαστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει αυτή την πρόταση αλλά να ζυγίσει καλύτερα την κατάσταση. Είναι πιστεύω πολύ σημαντικό να το έχω πει και αυτό και να το έχω βάλει στη συζήτηση. Ευχαριστώ η κυρία Σίπελ. Τελευταία. Ευχαριστώ πολύ, Κλοντ. Έχουμε 10 λεπτά επισήμω και δεν θα χρειαστώ και τα 10 λεπτά. Χαρά μου. Να προσθέσω κάτι. Υποστηρίζω σαφώς αυτά που είπε ο Μάικλ. Τα συζητήσαμε και στις συνεδρίες των συντονιστών. Το είπε και ο Τίμερμανς. Αν μιλάμε για δημοκρατία και για κράτος δικαίου, κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν μέσω αποφάσεων των δικαστηρίων και μέσω νόμων. Η δημοκρατία και το κράτος δικαίου όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ζούμε. Είναι βίωμα. Είναι το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Πώς εκτιμούμε την δημοκρατία. Πώς ενθαρρύνουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί τα δημοκρατικά του δικαιώματα το να υποστηρίζει κανείς τη δημοκρατία είναι και θέμα κοινωνικό. Αν αισθάνεται ο κόσμος ότι η ζωή του δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση, την πλειοψηφία, γιατί να ψηφίσουν. Και η ψηφοφορία είναι σημαντικότατο κομμάτι της δημοκρατίας. Καμιά φορά συμφωνώ. Δεν είναι μόνο φταίξιμο της κυβέρνησης. Χρειαζόμαστε ανεξάρτητα μέσα που μπορούν να ερευνούν και να ξεχνιάζουν υποθέσεις και κάποιες ΜΚΟ που έχουν τεχνογνωσία, εμπειρογνωμοσύνη να συμβουλεύουν, να παρουσιάζουν κάποια θέματα που ίσως να μας ξεφεύγουν στο πολιτικό μας έργο. Όμως υπάρχουν και κρίσιμα σημεία σε επίπεδο προσωπικού και ειδικών το έχουμε ξεκινήσει το θέμα, το συζητούμε. Πώς αποφασίζουμε ποια ΜΚΟ θα πάρει τα χρήματα, βάσει ποιων κριτηρίων. Ποιο μήνυμα θέλουμε να στείλουμε στα κράτη-μέλη, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ότι εμείς προσθέτουμε και συμπληρώνουμε μόνο κάτι, θα βρούμε λύση, είμαι σίγουρη. Διότι πρέπει να βρεθεί λύση. Ένα πρακτικό θέμα να τονίσω και ελπίζω να βρεθεί λύση γι' αυτό. Αν υπάρξει ένα νέο εργαλείο, ένα νέο μέσο και όχι υφιστάμενο που τροποποιείται για να προσαρμοστεί δεόντως. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Μια εποχή που πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι όχι μόνο λόγω Brexit ο προπολογισμό συρρυκνούται. Ξοδεύουν πολλά χρήματα σε αρκετά διαφορετικούς τομείς. Ελέγχοντας τα σύνορα για θέματα ασφαλείας και άμυνας σε όλα τα μέτρα ασφαλείας όπως τα στοιχεία επιβατών, τα PNR, ξοδεύουμε εκατομμύρια ευρώ και δεν έχουν καν υλοποιηθεί. Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα συνεχώς, αλλά παραμένει το, το σύνολο του υπολογισμού μικρό, παρά τις επιμέρους αυξήσεις. Δεν θέλω να απομακρυνθούμε από την ιδέα στήριξης των ΜΚΟ. Εγώ τι λέω να πιέσουμε περισσότερο τα κράτη-μέλη επί τη ευκαιρία αυτού είτε να δώσουν περισσότερα χρήματα για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό ή να έχουν άλλε ιδέε. Αυτό είναι θέμα τη Επιτροπή Λίμπε και λυπάμαι που το λέω πρόεδρε, είναι θέμα προπολογισμού. Είναι και θέμα ίσων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να γίνει κάτι στον τομέα των φόρων. Όλοι να καταβάλουν φόρους όλες οι επιχειρήσεις να πληρώνουν φόρους. Και ίσως μπορούμε να μιλήσουμε και για τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ούτως ώστε να έχουμε συμπληρωματικού πόρους. Αυτές είναι κάποιες ιδέες που θα συζητήσουμε. Η κεντρική ιδέα όμως να στηρίξουμε και τις ΜΚΟ είναι καλή. Υπήρξε και η ιδέα να σταματήσουμε κάποιες ΜΚΟ και αυτό ίσως είναι Ελπίζω μαζί να βρούμε όλοι τις δέουσες λύσεις. Ευχαριστώ. Καλώς. Ευχαριστώ, Μπίρκιτ. Για να είμαι ειλικρινής, αντικατοπτρίζεις τη θετική φύση της ιδέας, αλλά προβάλλεις και πόσο περίπλοκη είναι. Να πω το εξή. Οι συντονιστές το κατανόησαν. Έγινε μεγάλη προεργασία. Και ο κύριος Μπόνι συμμετείχε σε πολλές συναντήσεις και συζητήσεις και ταιριάζει με κάποιες σκέψεις άλλων συναδέλφων που εξέφρασαν διαφορετικές ιδέες επί διαφορετικής βάσης ενδεχομένω. Να πω το εξή λοιπόν. Περίπλοκο το θέμα, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Συμφωνούμε, βλέπετε, εν γέννη, τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να εξετάσουμε τον πολιτικό μηχανισμό, που είναι δημοσιονομικής φύσης. Είναι ένα ψήφισμα αυτό. Άρα σκιαγραφούμε τον πολιτικό μηχανισμό που συζητούμε. Αυτός είναι ο στόχος. Τον παρουσίασε ο κ. Μπόνι. Έγινε μία προετοιμασία συζήτησης, προετοιμασίας. Ας προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο ψήφισμα. Αυτό πιστεύω. Παρά τις ανησυχίες που εξέφρασε η Χέλγα και το ECR, οι ανησυχίες αυτές θα τροφοδοτήσουν και τις συζητήσεις για το ψήφισμα. Ήταν όμως απόφαση της πλειοψηφίας των συντονιστών να προχωρήσουμε προς το ψήφισμα και αυτό πρέπει να κάνουμε. Μίκαλ, γρήγορα, γρήγορα να κλείσουμε. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απόψεις σας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις καταστάσεις που είναι εναντίον της δημοκρατίας. Είμαστε, αυτό το θέμα είναι προς διάλογο, όχι για διαμάχη. Πρέπει να στηρίξουμε όλους τους φορείς εκείνους που είναι ανοιχτοί στο διάλογο και επιτρέπουν τη συμμετοχή πολλών ομάδων, επιχειρήσεων, φορέων, θεσμών, οργανώσεων. Συμφωνώ μετά με το πρόβλημα που παρουσιάστηκε από την Birgit. Είναι το πρόβλημα το οικονομικό του προπολογισμού. Αυτή είναι η ώρα που συζητούμε τον προπολογισμό. Άρα πρέπει να τεθεί το ζήτημα και μπορούμε να εγγυηθούμε στις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είμαστε ανοιχτοί προς συζήτηση. Πώς μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα μηχανισμό, να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει σαφήνεια περί λειτουργίας του μηχανισμού. Αυτή θα είναι η συνεισφορά μας. Όταν η πρόταση γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περαιτέρω συνεργασία προς εξέβρεση οθής βέλτιστης λύσης. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα εργαστούμε λοιπόν. Καλή δουλειά στο προσωπικό μας εύχομαι. Α, εσείς κάνετε, εσείς κάνετε τη δουλειά. Συγγνώμη, Δευτέρα Στρασβούργου βλέπετε. Ναι, βεβαίω ε, κάνετε τη δουλειά. Κάνετε τη δουλειά, Μπίρκετ. Σύντομο σχόλιο. Κοίτα, πράγματι, το είπα στο τέλος ότι είναι κάποια θέματα οικονομικά που τίθενται, αλλά εγώ αισθάνομαι υπεύθυνη γιατί στο τέλος τα χρήματα από κάπου πρέπει να έρθουν. Και ό,τι αποφασίσουμε εμείς είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Λοιπόν, ήθελα απλώ να αναφέρω ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι ίσω υπάρξουν κάποια προβλήματα. Και δεν θα ήμουν ικανοποιημένη αν έχουμε χρηματοδότηση για τις ΜΚΟ και πάρουμε χρήματα από άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν άλλη επιτροπή, όπως τη ΛΥΜΠΕ. Ας σταματήσουμε όμως εδώ. Στο ψήφισμα μπορούμε να το καλύψουμε αυτό. Έχουμε καλύψει πολύ πιο περίπλοκα ζητήματα. Είπε τρέφοντας ελπίδες ο μιλητής. Λοιπόν, Προσβλέπουμε συνεδρίαση της ομάδας, σχετικές συζητήσεις. Πείτε μου πότε θα διεξαχθούν, για να μην παρίσταμε σε αυτές. Μίκελ, το ξέρεις θα έρθω, θα έρθω. Αν με χρειαστείς εκεί θα είμαι. Καλή τύχη. Αλλά είναι περιθώριο στενό το χρονικό. Θα το κάνω όμως συμφωνήσαμε. Καλή τύχη. Συνάδελφοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σήμερα, Δευτέρα Στρασβούργου. Το εκτιμώ, το εκτιμώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Πέρα συνεδριάσεως. Καλό βράδυ και πάλι.